συνάδελφοι και καλεσμένοι. Είμαι ο Πρόεδρος και με μεγάλη μου τιμή ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική θητεία να σας καλωσορίσω στην ακρόαση αυτή. Αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε αυτό το εργαστήριο για να συζητήσουμε για το μέλλον του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρόντες ομιλητές, καθώς και το Policy Department που οργάνωσε αυτό το εργαστήριο εκ μέρους της Επιτροπής μας. Θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει ένα ρόλο να παίξει, όχι μόνο στην οικοδόμηση του δικαίου, αλλά συμμετέχει και σε διάφορες νομοθετικές διαδικασίες και στην προώθηση του νομικού σώματος εν το συνόλο του. Τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει για αυτό το εργαστήρι θα πρέπει να τα δείτε ως σημάδι και απόδειξη αυτής της συμμετοχής μας. Πέντε θέματα έχουμε επιλέξει που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά διαφόρων δυνατοτήτων ε, ανάπτυξης του ευρωπαϊκού δικαίου. Καταρχάς, θα ακούσουμε την εμπειρία του δικαστηρίου για, από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε εθνικό επίπεδο τα εθνικά σας δικαστήρια ε, εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο και είναι τμήμα αυτού. Και επομένω ε, παίρνουν αποφάσει για κάθε λογή θέματα. Συν το χρόνο, η θέση του ευρωπαϊκού δικαίου φυσικά έχει αλλάξει και οι εθνικοί δικαστέ είναι πολύ πιο άνετοι με την ιδέα εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και το σώμα του ευρωπαϊκού δικαίου έχει βεβαίω αυξηθεί ποσοτικά και ελπίζουμε και ποιοτικά. Οι δύο μας ομιλητές θα μας μιλήσουν για την άποψή τους από αυτή τη Δεύτερον, θα ξέρετε ότι η Επιτροπή μας έχει την κύρια ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και εκδίδει και μία αιτήσια έκθεση γι' αυτό. Ο κύριος Μπαλέστερος θα σας μιλήσει για τους προβληματισμούς του, για το πώς θα καταστήσουμε αποτελεσματική αυτή την παρακολούθηση, αυτό το monitoring του Κοινοβουλίου. Θα ακούσουμε επίσης μια παρουσίαση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Είχαμε ακούσει τον καθηγητή Κράμερ πολλές φορές στο παρελθόν για αυτό το θέμα, την καθηγήτρια μάλλον, και πιστεύουμε ότι οι απόψεις της θα ενδιαφέρουν πολύ την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται πολύ για περιπτώσεις όπου οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων της δικαιοσύνης πρέπει να συμπληρωθούν. Έχουμε δύο ε, εμπειρογνώμονες που θα μας μιλήσουν για τις μελλοντικέ πιθανές εξελίξεις ε, του ευρωπαϊκού ε, δικαίου στην πνευματική διοκτησία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε εξελίξεις. Έχουμε το, την Ευρωπαϊκή ευρυστεχνία και, για το, και το δίκαιο για το εμπορικό σήμα και θα ακούσουμε και εμπειρογνώμονες επίσης από την Σκόλα Superiore, την ανώτατη σχολή Σαντάνα στην Ιταλία, που θα συζητήσουν για ένα τελείως νέο τομέα δικαίου, που ασχολείται με τη ρομποτική και τα αυτοματοποιημένα συστήματα και το σχετικό δίκαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το, να απαντηθεί το ερώτημα ποιο είναι νομικά υπεύθυνο για μια απόφαση που λαμβάνει ένα ρομπότ. Ανάμεσα στις παρουσιάσεις και μετά τις παρουσιάσεις θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι κάθε ομιλητής θα παρουσιάσει την παρουσίασή του και για αυτή την παρουσίαση υπάρχει και γραπτή ομιλία που υπάρχει και σε υπόθεμα χαρτιού, αλλά και στην ιστοσελίδα. Θα ακούσουμε καταρχάς τον ε, πρώτο μας ομιλητή, τον Wolfgang Χόιζελ, που είναι Διευθυντής της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ε, κύριε Χόιζελ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας, για την ε, εισαγωγή σας, τα ευγενικά σας λόγια. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τα μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα παρά τα αγγλικά. Φυσικά έχω τη δυνατότητα να σας απαντήσω και στα αγγλικά αν χρειαστεί ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή να σας ε, μιλάω σήμερα για ένα θέμα το οποίο είναι κάπως ε, βαρετό ίσως για το ρόλο και την ευθύνη του Εθνικού Δικαστή στην εφαρμογή του Εθνικού Δικαίου ένα θέμα το οποίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια κοινότητα δικαίου και βασίζεται στο δίκαιο, είναι βεβαίως πάρα πολύ ουσιαστικό και ε, μας απασχολεί. Οπότε το θέμα εδώ πέρα δεν είναι οι μελλοντικέ εξελίξεις, είναι οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη χρήση και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ρόλο έχει ο Εθνικός Δικαστής στην εφαρμογή αυτή. Εγώ είχα κάνει κάπως διαφορετικό τίτλο. Το θέμα δεν είναι εμπειρίες στην αίθουσα του αλλά για την εφαρμογή του δικαίου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Δεν είναι εμπειρική η μελέτη μας, δεν είχαμε χρόνο και δυνατότητα. Η πρόκληση που ε, αποτελεί αυτό νομίζω φαίνεται με το να παρουσιάσω τις ε, διάφορες διαδικασίες ε, που πρέπει να γνωρίζει ο εθνικός δικαστής θα αναφερθώ σε κάποιες ε, βασικές ε, αρχές αλλά βεβαίως ε, και την διαδικασία της προδικαστικής απόφασης η οποία θα έλεγα ρυθμίζει και κανονίζει έναν θεσμικό διάλογο μεταξύ του Εθνικού Δικαστή και του ΔΕΚ. Πρέπει λοιπόν σήμερα ο Εθνικός Δικαστής να ξέρει κάποια πράγματα για τα μέσα αυτά της ε, δικαστικής συνεργασίας. Το, πιστικό και το, το ποινικό με και δίκαιο έχουν πάρα πολλές ε, δυνατότητες ε, αλλά βεβαίως θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Όλα αυτά βεβαίως με οδηγούν στο να πω πως βεβαίως όλες αυτές οι γνώσεις και οι ικανότητες ε, του δικαστή όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου θα έχουν πραγματικά ε, επίδραση και εφαρμογή μόνο αν υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και μάλιστα σε εθνικό ε, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για εμένα. Είμαι διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Ακαδημίας ε, Δικαίου που ιδρύθηκε το 1992 μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς εν ώψη της ε, ενιαίας αγοράς. Το 1992 δηλαδή γνώριζαν οι πολιτικοί πως με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα έπρεπε οι δικηγόροι και οι δικαστές στο εθνικό δίκαιο να αναλάβουν νέες ευθύνες ε, ε, και μέχρι τότε πρακτικά δεν ήξεραν τίποτα για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εγώ προσωπικά ήμουν δικαστής ε, τότε στην Γερμανία και η εμπειρία μου τότε ήταν ότι αποφεύγαμε την επαφή και τα ερωτήματα προς το 10 το πολύ πολύ αναγνωρίζαμε πως ε, ήταν, ένα ήταν ε, θέματα που έπρεπε να επιληφθούν από ε, άλλα δικαστήρια σε υψηλότερο βαθμό. Θα ήθελα να πω πως α, όσον αφορά τον ρόλο του Εθνικού Δικαστή βλέπουμε εδώ πέρα πως υπάρχουν δύο προκλήσεις. Το ένα είναι η πρόκληση για τον ίδιο τον Εθνικό Δικαστή, ο οποίος ήδη σήμερα από την εκπαίδευσή του δεν εκπαιδεύεται κατά κύριο λόγο ως χρήστης και ο κάποιος ο οποίος θα εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Από την άλλη, ε, υπάρχει ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, μιλάει για μια ενιαία εφαρμογή, αλλά από ό,τι φαίνεται επαφίεται σε μια αποκεντρωμένη ε, πρακτική. Και βλέπουμε επίσης πως το ευρωπαϊκό δίκαιο συνεχώς ε, αυξάνεται και όσον αφορά το πεδίο του, αλλά και όσον αφορά την πολυπλοκότητα. Για να μπορέσει λοιπόν ο Εθνικός Δικαστής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το μεγαλύτερο όγκο και έκταση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και να το εφαρμόσει, ήδη από πάρα πολύ νωρίς, τη δεκαετία του 60, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε δύο αρχές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Εθνικός ε, Δικαστής. Έχουμε δηλαδή την αρχή του ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται ε, άμεσα και αφετέρου έχουμε την αρχή της ε, υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού. Αρχές οι οποίες έχουν ε, τονιστεί επανειλημμένα και εξελιχθεί από την ομολογία του ΔΕΚ και Βεβαίως ε, αυτό το αναγνωρίζουν και τα εθνικά δικαστήρια ε, γιατί βλέπουν πως όταν υπάρχει μια σύγκρουση πράγματι αναγνωρίζουν ε, πως κατησχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και βεβαίως αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, κάποιο ερώτημα, υπάρχει ακριβώς αυτή η διαδικασία της παδικαστικής απόφασης όπου τίθεται το ζήτημα ε, του πώς και ποιος ε, μπορεί να λάβει μία απόφαση. Η Ακαδημία μας είχε, κάνει, είχε αναλάβει την ευθύνη να κάνει μία μελέτη για την εκπαίδευση των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό ε, δίκαιο. και είχαμε διαπιστώσει πως ειδικά στον τομέα αυτών των προδικαστικών ερωτημάτων δεν ξέρουν πως λειτουργεί η διαδικασία, οι εθνικοί δικαστές γνωρίζουν ότι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, αλλά κατά κανόνα δεν την έχουν χρησιμοποιήσει. Οπότε εδώ πέρα ε, πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση. Επίσης βλέπουμε πως με την εξέλιξη του κεκτημένου στον τομέα της ε, δικαιοσύνης, ε, παραδείγματο χάρη στο ποινικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο, έχουμε νέες ε, διαδικασίες, την επιταχυμένη διαδικασία συγκεκριμένα στα προδικαστικά ερωτήματα και μάλιστα τι γίνεται, παροτρύνεται ο δικαστής να προτείνει ο ίδιος μία απάντηση στην ερώτηση στην οποία στέλνει στο ΔΕΚ. Δύο λόγια τώρα για το θέμα εκείνο το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα από το συνθήκη του Άμστερνταμ και εδώ δηλαδή την ε, συνεργασία και σε ποινικά και σε αστικά θέματα από την Σύνοδο Κορυφής του Τάμπερε με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δικαστηρίων και έχει εφαρμοστεί με διάφορα μέσα στην πράξη και νομίζω έχει αποδείξει πως λειτουργεί και βεβαίως αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να διατάξουμε. Είναι κάτι το οποίο θα αναπτυχθεί όταν γνωρίζουν οι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη ποια είναι η ανταπόκριση από τις άλλες χώρες και όταν έχουν πιστεί πως ε, πράγματι εφαρμόζονται οι ίδιες ε, αρχές όπως και στη χώρα τους. Γνωρίζετε πως ε, το πρόγραμμα αυτό του Τάμπερε και της Στοκχόλμης προωθήθηκε με πενταετή προγράμματα και δημιουργήθηκαν έτσι και τα κατάλληλα πλαίσια. Από τον Ιούλιο 2014 έχουμε και τη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας και έχουμε πλέον στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Και Ε, κύριο στόχο έχουν ε, την ε, κωδικοποίηση πλέον. Δηλαδή το μεγάλο ερώτημα είναι πού θα πάμε όσον αφορά την κωδικοποίηση αυτών των μέσων. Είναι λογικότερο να πάμε προς την κατεύθυνση των διαφόρων αστικών νομοθετημάτων ή και ποινικών νομοθετημάτων που είναι διασπαρμένα παντού. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έχει αποφασιστική σημασία το πώς θα απαντηθεί και θα οδηγηθούμε πιθανώς σε νέες ε, νομοθετικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία στο πεδίο του αστικού δικαίου θα ήθελα να αναφέρω το τι περιέχεται στο εγγραφό μας. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ερωτημάτων περί αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ήδη από το 1986 υπήρχε μια σχετική συμφωνία, πριν δηλαδή από, το, από την ε, ε, σύσταση του χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης και βεβαίω είχε αναγνωριστεί πως είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο εάν θέλουμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά. Υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα στον ε, τομέα αυτό μια συνεχής εξέλιξη και είναι σαφές πως οι εθνικοί δικαστές οι οποίοι πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα τον κανονισμό αυτό σε περιπτώσεις διασυνοριακής αρμοδιότητας ή εκτέλεσης απόφασης πρέπει να γνωρίζουν πώς λειτουργεί το ίδιο και στον τομέα της ε, χρεοκοπίας ε, το οποίο μπορεί να αφορά παραδείγματος χάρη έναν όμιλο επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες και εκεί πέρα υπάρχουν σοβαρές απαιτήσει από τους δικαστές και υπάρχει και ο τομέας του οικογενειακού δικαίου και ενδιαφέρουν οι διασυνοριακές περιπτώσεις διαζυγίου, διατροφής κτλ. Από την άλλη βλέπουμε πως υπάρχει ο τομέας της ε, ποινική ε, συνεργασίας όπου ήδη εδώ και ένα χρόνο υπάρχει η πρόταση της Κομισιόν για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία, ε, η οποία θα ασχολείται πρώτα απ' όλα με την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα έχει οπωσδήποτε την δυνατότητα να ασχολείται με διασυνοριακά εγκλήματα. Το γνωστότερο τέτοιο παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, Και μην ξεχνάμε πως πράγματι εδώ πέρα υπάρχει σοβαρή κριτική στην πράξη, π.χ. το ότι κάποιες χώρες ε, το χρησιμοποιούν δυσανάλογα ή η διαδικασία για τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι πάρα πολύ πρακτική και δεν υπάρχει μία ενιαία πρακτική. Και επειδή βεβαίως ε, είναι ένα σύστημα διακυβερνητικό δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η μεγάλη τυποποίηση στην εφαρμογή του. Αυτά για τα ουσιαστικά θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο Εθνικός Δικαστής ε, και τις ικανότητε πρέπει να έχει για να τα διαχειριστεί. Αυτό το οποίο δεν ανέφερα καθόλου βεβαίως είναι το θέμα της διασυνοριακής εφαρμογής, δηλαδή ποιο εθνικό δίκαιο ισχύει σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση, αλλά και βεβαίως ε, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο εθνικός δικαστής και εάν ε, εφαρμόζει κάποιο ξένο, κάποια ξένη νομιτάξη πρέπει να ξέρει τι ισχύει σε αυτήν. Οπότε θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ στο θέμα της ε, μετεκπαίδευσης. Είναι σαφές ε, πως η μετεκπαίδευση στη δικαιοσύνη είναι πρώτα απ' όλα αποστολή των εθνικών διοικήσεων και των σχολών δικαστών. Αλλά νομίζω είναι επίσης σαφές πως υπάρχει μεγάλη ευθύνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει μια αρμοδιότητα θα έλεγα για την υποστήριξη αυτής της εκπαίδευσης και πρέπει να το δούμε αυτό ευρεία τη ενία. Δηλαδή να μην περιοριστούμε μόνο στους δικαστές αλλά πιθανώς και στους δικηγόρους. Πιθανώς ο δικηγόρος είναι αυτός ο οποίος πρώτος θα έρθει αντιμέτωπος με μια υπόθεση και θα διαπιστώσει πως έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much, uh, Dr. Σας ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρα Χόιζελ για την εκτενή σας εισήγηση. Μας μιλήσατε για όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου που θα πρέπει να λάβει υπόψη ο εθνικός δικαστής μέσα στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός του ή τη. Ε, συνέβη ένα θαύμα. Ήδη μετά το δεύτερο σημείο προτρέχουμε του προγράμματος. Είμαστε πολύ καλά από πλευράς ώρας, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Η δεύτερη ομιλήτρια, ή, μάλλον είναι ο ε, καθηγητής Στότς, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είμαι Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Ε, σας ε, εύχεται κάθε επιτυχία στη διάσκεψη αυτή. Το θέμα που σας απασχολεί δηλαδή η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά δικαστήρια αποτελεί, έχει μάλλον μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μέσω του ε, προδικαστικού ερωτήματος, δυνάμει του άρθρου 267, ε, λαμβάνουμε υπόψη την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από το εθνικό ή όπως ορίζει το δικαστήριο. Δυνάμει του άρθρου 267 προβλέπεται μία συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Εθνικών Δικαστηρίων όπου τα εθνικά δικαστήρια θέλουν και επιδιώκουν την σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Στην εισήγησή μου θα ήθελα να προβώ σε ορισμένα γενικά σχόλια σε σχέση με το προδικαστικό ερώτημα δυνάμει των συνθήκων. Για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή αυτή, το προδικαστικό ερώτημα, ε, κατέχει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο στις διαδικασίες του και Μεταξύ 2009 και 2013 οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυξήθηκαν κατά 20%. Δηλαδή από 590 υποθέσεις φτάσαμε σε 700 και τα προδικαστικά ερωτήματα έχουν αυξηθεί κατά 60% από 500, 259 το 2009 ε, πέρασαν σε 413 το 2013. Το 2009 τα προδικαστικά ερωτήματα ήταν το 45% του δικαιοδοτικού έργου, ενώ το 13 αποτελούν το 60% της δραστηριότητας του δικαστηρίου. Αυτά τα στοιχεία ε, δεν... Μάλλον δεν έχουμε πλήρη στοιχεία για το 14. Είχα, 242 προδικαστικά ερωτήματα μέχρι τώρα που αποτελούν το 71% της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του δικαστηρίου. Δηλαδή πάνω από το 2 τρίτα των ε, υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου. Ερωτήματα που προέρχονται από τα εθνικά δικαστήρια. Σχετίζονται με διάφορα θέματα αλλά σχετίζονται ιδιαίτερα με τον χώρο της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ε, την προστασία των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Ως προς την κατανομή των προδικαστικών ερωτημάτων ε, μπορούμε να πούμε ότι οι Γερμανοί δικαστές ε, υποβάλλουν τα περισσότερα ερωτήματα. 21,5% των προδικαστικών ερωτημάτων το 2013 και στη συνέχεια έρχονται οι Ιταλοί 13,7%, ο Ολλανδοί 9,7%, 5,7% οι Βέλγοι και οι Γάλλοι με 5,3%. Για τα 10 κράτη-μέλη που προσχώρησαν το 2014, η ποσοστή αναλογία το 2013 ανέρχεται σε 15% για τη Ρουμανία, 3,5% και για τη Βουλγαρία 2,22%. Τέλος, στις 26 Μαΐου του τρέχοντος τα πρώτα προδικαστικά ερωτήματα υποβλήθηκαν από τις κροατικές δικαστικές αρχές σε σχέση με το δίκαιο του περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, το Σεπτέμβριο του 2012 ε, ένας νέος ε, ε, κανονισμός ετέθησε ισχύ στο δικαστήριο που λαμβάνει υπόψη αυτή την εξέλιξη και τα προδικαστικά ερωτήματα εντάσσονται σε αυτό το νέο κανονισμό και ο πρόεδρος του δικαστηρίου μίλησε για τους ε, βασικούς στόχους του κανονισμού έτσι ώστε να υπάρξει μια συνέχεια με τον παλαιό κανονισμό για να προσδοθεί μεγαλύτερη σημασία στα ε, προδικαστικά ερωτήματα με μείωση της ε, διαδικασίας. Ως προς το τελευταίο αυτό ζήτημα, το διάστημα λήψης αποφάσεων περάσαμε από 23 ε, μήνες το 2004 σε 17 μήνες το 2009 και σε 16,3 μήνες το 2013. Τα αριθμητικά στοιχεία για το 2014 είναι ακόμα καλύτερα. Εάν πρόκειται για επίγον προδικαστικό ερώτημα, σε ορισμένες περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να δικάσει κατά προτεραιότητα, να εκδικάσει κατά προτεραιότητα. Πρόκειται για υποθέσεις επίγοντος χαρακτήρα και η απόφαση λαμβάνεται μεταξύ 6 και 8 εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση κάθε χρόνο εκδικάζονται δύο με, τέσσερις, με τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα ε, ετησίως. Ε, στα πλαίσια του προδικαστικού ερωτήματος ε, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και θα πρέπει να σταθώ σε δύο ζητήματα. Πρόκειται για δύο σχόλια ως προς τη διαδικασία και ως προς την ουσία, δηλαδή την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Σε σχέση με το διαδικαστικό σκέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το μη παραδεκτό, την μη αποδοχή, μάλλον το μη παραδεκτό ή παραδεκτό των ε, προδικαστικών ερωτημάτων. Το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού προβλέπει ότι όταν το δικαστήριο κρίνει αυτό αναρμόδιο για να εκδικάσει μία περίπτωση, τότε απορρίπτεται η προσφυγή και ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει να ε, δώσει ε, τέλος αυτή τη διαδικασία τα ερωτήματα σε σχέση με την αρμοδιότητα του δικαστηρίου και ως προς το παραδεκτό ε, κρίνονται αυτεπαγγέλτος από τον Ευρωπαίο Δικαστή. Σύμφωνα με την ε, πάγια νομολογία του δικαστηρίου, στα πλαίσια ενός προδικαστικού ερωτήματος, δυνάμει του άρθρου 267 το δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει το κοινοτικό δίκαιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Το ίδιο ισχύει και για τα προδικαστικά ε, ερωτήματα ε, τα οποία ε, κρίνονται προδικαστικά καθαρά. Ο Εθνικός Δικαστής υποβάλλει ένα ερώτημα ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κατά πόσο μια εθνική ε, διάταξη είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο για να ερμηνεύσει το εθνικό δίκαιο καθεαυτό. Το δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει αποκλειστικά το κοινοτικό δίκαιο. Άρα είναι αναρμόδιο να κρίνει εθνικά, το, το εθνικό δίκαιο. Άρα μπορεί να κρίνει κατά πόσο είναι συμβατή μια εθνική διάταξη με το κοινοτικό δίκαιο. Αντί να απορριφθεί το ερώτημα ε, λόγω αναρμοδιότητας, το δικαστήριο μπορεί να το επαναδιατυπώσει δίδοντας τα ε, στοιχεία ερμηνείας στο Εθνικό Δικαστήριο για να μπορέσει να κρίνει την συμβατότητα του, των εθνικών διατάξεων με το κοινοτικό δίκαιο. Δηλαδή το ερώτημα του Εθνικού Δικαστή δεν κρίνεται ε, μη παραδεκτό και το ε, δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί επαναδιατυπώνοντας ε, το ερώτημα. Επειδή έχω εργαστεί και στο γραφείο ενός δικαστή, μπορώ να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εθνικοί δικαστές προβαίνουν σε ένα λάθος διατύπωσης, χωρίς βεβαίως σοβαρές συνέπειες. Το Δεύτερο σκέλος αφορά την αρμοδιότητα όπου μιλάμε για καθαρά εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή κατά πόσο τα στοιχεία της κύριας δίκης ε, αφορούν αποκλειστικά ένα κράτος μέλος. Ε, πρόσφατα το δικαστήριο έκρινε αυτό αναρμόδιο να αποφανθεί ε, σε σχέση με ένα βουλγαρικό ερώτημα για μία εντολή σύλληψης με βάση έναν έλεγχο που διενεργήθηκε σε βουλγαρικό έδαφος ενός πολίτη ο οποίος ε, δεν παρουσίασε την εθνική του ταυτότητα. Δηλαδή όταν πρόκειται για καθαρά εθνικά ζητήματα, το δικαστήριο κρίνει αυτό αναρμόδιο διότι δεν μπορεί να αναμειχθεί με το εθνικό δίκαιο αλλά δεν είναι όλες οι υποθέσεις τόσο προφανείς. Σε μια άλλη υπόθεση, σε σχέση με την υποχρέωση των γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά ορισμένων ασθενειών, το ανώτατο Σλοβακικό Δικαστήριο υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ σε σχέση με, την υποχρεωτική, με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό διότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να ε, εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη και το ενωσιακό δίκαιο. Το δικαστήριο αυτό ρώτησε εάν το άρθρο 188 της Συνθήκης για την αρμοδιότητα της Ένωσης στα θέματα δημόσιας υγείας θα πρέπει να ερμηνευθεί ε, υπό την έννοια ότι οι στόχοι που πρέπει να ε, υλοποιήσουμε σε ό,τι αφορά την πρόληψη των ασθενειών δεν επιτρέπουν σε έναν πολίτη της Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρνηθεί υποχρεωτικό εμβολιασμό. Το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι το άρθρο αυτό της συνθήκης δεν επιβάλλει υποχρεώσει στα κράτη των ανηλίκων που θα μπορούσαν να προταθούν για να ε, κριθούν τα εθνικά μέτρα κατά πόσο είναι σύμμορφα. Ε, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι εντελώ αναρμόδιο το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή για να αποφασίσει για τέτοιου τύπου θέματα. Πρόεδρε, τα θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου ε, αποτελούν αντικείμενο εντελώ προκαταρτική εξέτασης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι αρμόδιο για να απαντήσει σε ένα τέτοιο τύπου ερώτημα, τότε απορρίπτει το αίτημα. Και το αναπέμπει στην εθνική δικαιοσύνη για λόγους έλλειψης αρμοδιότητας. Δεύτερη παρατήρηση διαδικαστικής φύσεως αφορά ένα άλλο άρθρο του καονισμού διαδικασιών που είναι το άρθρο 94, όπου για πρώτη φορά ο καονισμός για τα διαδικαστικά μιλάει για κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται, ούτω ώστε μια εθνική, ένα εθνικό αίτημα από εθνικό δικαστή να γίνει παραδεκτό. Ε, θα πρέπει να εξηγηθεί συνοπτικά ε, η διαφορά, θα πρέπει να αναφερθούν τα γεγονότα, δεύτερον, όπως ε, τα αντιλαμβάνεται το δικαστήριο. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές διατάξεις για αυτή την περίπτωση και αν χρειάζεται το εθνικό δικαστήριο πώς τα εξηγεί. Και τρίτον να ε, υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη που να δικαιολογεί γιατί ζητάει μια ερμηνεία ε, των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω τι είπε ο καθηγητής Χόισελ. Φυσικά οι δικαστές υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούν αυτό το δικαίωμα παραπομπής του ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καθώς και τις απαιτήσει από το νέο κανονισμό, το διαδικαστικό. Θα ήταν ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει στο, στην ιστοσελίδα του δημοσιεύσει συστάσεις, να σας αναφέρω κάποια έγγραφα ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασέλιδο είναι αυτό, ε, προς τα εθνικά δικαστήρια που αφορά την εισαγωγή προδικαστικών διαδικασιών. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το έγγραφο που κάθε εθνικός δικαστής θα πρέπει να συμβουλεύεται πριν παραπέμψει μία υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν οι παραπομπές αυτές δεν σέβονται τις τυπικές αυτές προϋποθέσεις, τότε το δικαστήριο τι ακυρώνει, δεν τις δέχεται, γιατί τις κρίνει μη παραδεκτές. Θα πρέπει το δικαστήριο λοιπόν να ενημερώνεται πολύ καλά γύρω από το πλαίσιο και τα γεγονότα που αιτιολογούν αυτό το αίτημα του Εθνικού Δικαστή. Γι' αυτό λοιπόν ο εθνικό δικαστή θα πρέπει να σέβεται όλα αυτά τα στοιχεία, τα τυπικά δηλαδή, τι τυπικές προποθέσει. οι περιπτώσεις όπου απορρίπτει ένα ερώτημα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί το θεωρεί μη παραδεκτό ή θεωρεί αυτόν ε, αναρμόδιο, αποτελούν το 6% του συνόλου των αιτήσεων. Δεν είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αμεληταίο. Τελευταία ερώτηση. Και θα περιοριστώ εδώ γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει. Το θέμα της ε, εφαρμογής του, χα της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Η Χάρτα εφαρμόζεται 100% σε ό,τι αφορά το παράγωγο δίκαιο. Δηλαδή το δίκαιο το οποίο απορρέει και παράγεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή της χάρτας ε, σε εθνικό επίπεδο, το άρθρο 51.1 των θεμελιωδών δικαιωμάτων λέει ότι ο χάρτης ε, εφαρμόζεται αποκλειστικά στο βαθμό που το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο. Εφαρμόζεται. Έχουμε μία ε, απόφαση του 2013 όπου το δικαστήριο διευκρίνησε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται η χάρτα σε εθνικό επίπεδο και είπε πολύ ξεκάθαρα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυάται η χάρτα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν μια εθνική νομοθεσία ε, υπησέρχεται στο πεδίο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη ε, συνάφεια με την εφαρμογή του παράγωγου δικαίου που θα πρέπει να σεβαστούν τα κράτη-μέλη και την εφαρμογή της χάρτας σε εθνικό επίπεδο. θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια της ένομης τάξης. Και είναι εύκολο να εφαρμοστεί αυτό από τους εθνικούς δικαστές. Όταν τα δικαστήρια, ε, ή μάλλον όταν τα κράτη λειτουργούν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων, τότε είμαστε εκτός του πεδίου εφαρμογή του δικαίου τη ε, Ένωση, τότε ο χάρτη δεν εφαρμόζεται. Στην αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται. Υπάρχουν διάφοροι συγγραφεί οι οποίοι αμφισβήτησαν αυτή την ομολογία. Και υπάρχουν και κάποια δικαστήρια μάλιστα τα οποία έχουν εκφράσει κάποιες αμφιβολίες. Αλλά εδώ μπορούμε να πούμε το εξή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε αντίθεση με τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, και σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου δεν είναι μια εξειδικευμένη, ένα εξειδικευμένο δικαστήριο που ασχολείται αποκλειστικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του, του Λουξεμβούργου είναι πολύ πιο ευρεία. Ε, ερμηνεύει το σύνολο του ενωσιακού δικαίου και καλύπτει πάρα πολλού τομεί. Και ακριβώ ε, παγρυπνεί ούτω ώστε και στην περίπτωση τη χάρτα να μην υπάρχει ανταγωνισμό ανάμεσα ε, στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στο ρόλο άλλων δικαστηρίων που είναι εξειδικευμένα για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, Πρόεδρε, και είμαι τώρα έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον καθηγητή Στότς. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Πριν να ανοίξουμε τη συζήτηση. Έχουμε μάλλον ακόμα μία ομιλήτρια, την κυρία Μάρτα Μπαρλέστέρος, που θα μιλήσει και αυτή και μετά θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές για ερωτήσεις. Γεια σας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτό το εργαστήριο. Λέγομαι Μάρτα Μπαγέστερος από ένα γραφείο συμβούλων που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών για θέματα πολιτικής στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για περιβαλλοντικά θέματα, ε, θέματα υγείας καταναλωτών, ε, Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα κάνω μια εισαγωγή με κάποιες διευκρινήσεις για κάποιους όρους που χρησιμοποιούμε και εν συνεχεία θα μιλήσω για την ε, μεταγραφή του ανοσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση και τέλος τα εργαλεία ε, εφαρμογής καθώς και τις διαδικασίες ε, σε περίπτωση παραβάσης, παράβασης. Θα ήθελα να σας τονίσω καταρχήν ότι αυτή η ομιλία που την έχετε και στην ιστοσελίδα αλλά και σε φυλάδια θέλει να τονίσει την ανάγκη για ισχυρές ε, ενωσιακές πολιτικές για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε εθνικό επίπεδο. Οι προηγούμενοι ομιλητέ μίλησαν για αυτό το επίπεδο. Εγώ θέλω να μιλήσω για το ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα. Για το επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Εδώ μιλάμε για τι δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώ και τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συνήθω, και θα ήθελα να διευκρινίσω, έχουν την μετεγγραφή, transposition, που αναφέρεται σε νομικές πράξεις που θα χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να ενσωματωθεί η ενωσιακή νομοθεσία στο ε, εθνικό, στην εθνική τάξη. Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αφορά το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία στην πράξη στα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή αναφέρεται και στα δύο, και στην μετεγραφή και στην εφαρμογή. Και η enforcement, το enforcement αφορά τα μέτρα που υιοθετούνται από τις δημόσιες αρχές για να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση και την εφαρμογή του, ε, του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή α, μεταγραφή και εν συνεχεία χρήση και ενσωμάτωση, ας πούμε, και εφαρμογή. Λοιπόν, ποια είναι τα πόρισματα της μελέτης μας. Είναι κυρίως δύο. Να σας τα πω γενικά και θα μπω σε λεπτομέρειες. Γενικά, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα μακρόπνο πρόβλημα με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και η Κομισιόν επομένως δυσκολεύεται στην, να εξασφαλίσει μια συστηματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Έχει δυσκολία να εντοπίσει και τις παραβάσεις, αλλά και να εξασφαλίσει τον έλεγχο όλων των παραβάσεων. Και για αυτό το λόγο θα μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Κομισιόν, ούτω ώστε να παίξει σωστά αυτό το ρόλο. Για την μεταγραφή, transposition, η Κομισιόν παρακολουθεί την έγκαιρη μεταγραφή και σωστή μεταγραφή των οδηγιών και αυτή είναι μια προτεραιότητα που αναγνωρίζεται σε διάφορα έγγραφα, αλλά κυρίως στις διάφορες αιτήσεις εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου που δημοσιεύονται ετήσια. Υπάρχει μια γενική τάση στη μεταγραφή ή μεταφορά να υπάρχει καθυστέρηση από τα κράτη-μέλη στην μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στην Εθνική Ενωμή Τάξη. Αναγνωρίζεται αυτό στην τελευταία ετήσια έκθεση που μιλάει για το 2012, όπου λέει ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη είχαν ε, υποστεί διαδικασίες επί παραβάση. Παραδείγματο χάρη. Ε, η οδηγία που μιλάει για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κρατών μελών. 24 κρατημέλη είχαν υποβληθεί σε τέτοιε διαδικασίε επί παραβάση. Ε, έχει αυξηθεί η... Έχουν αυξηθεί οι παραβάσει δηλαδή, οι οποίες, και οι διαδικασίε επί παραβάση που ξεκίνησε η Κομισιόν από το 2009 στο 2011. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν δηλώνει Συζητώντα με τα κρατη ότι η επίπτωση του άρθρου 260 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 263, ε, είχε σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ε, μεταφοράς και εφαρμογής στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Όταν ξέρουν τα κρατημέλη ότι θα υποστούν τέτοιε διαδικασίε επιβαραβάση, ε, αντιδρούν πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτό το άρθρο λοιπόν ε, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμα στα κράτη-μέλη για την καθυστερημένη μεταφορά από την πρώτη στιγμή που φτάνουν αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Δεν χρειάζεται δηλαδή ε, να υπάρξει δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου. Ήδη από την πρώτη φορά επιβάλλονται πρόστιμα. Και η αποτελεσματικότητα αυτού του άρθρου έχει αυξηθεί το... Έχει αυξήσει μάλλον το επίπεδο μεταφορά τη ανοσιακής νομοθεσία στην Εθνική νομητάξη. Τάξη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αποφασιστεί ότι όντω υπάρχει παράβαση. Τα βασικά φράγματα για την έγκαιρη και σωστή μεταφορά έχουν εντοπιστεί ως ε, η αοριστία των οδηγιών πρώτον και αυτό είναι και αυτό οφείλεται σε πολιτικούς συμβιβασμούς κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Δηλαδή, θα θέλαμε εδώ να θέσουμε υπόψη του Κοινοβουλίου το εξή θέμα. Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, καλό είναι να προκύπτουν νομοθεσίες ακριβής εναργής. Επιπλέον, υπάρχει ένα πρόβλημα σε επίπεδο κρατών μελών, όπου έχουμε διαφορετικές θεσμικές διαδικασίες που υπάρχουν για την υιοθέτηση της, και εφαρμογή της μεταφερόμενης νομοθεσίας. Δηλαδή, προς αυτήν την κατεύθυνση τώρα πιστεύουμε ότι οι συστάσεις για την βελτίωση της μεταφοράς υπάρχουν για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα κρατημέλη έχουν δημιουργήσει τις σωστές δομές για να εξασφαλίσουν ότι το άτομο που διαπραγματεύεται κατά διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας το συγκεκριμένο μέτρο, όταν ας πούμε διαπραγματεύεται την οδηγία, είναι σε επαφή με τους ανθρώπους που θα εφαρμόσουν μετά αυτή την οδηγία. Θα τη μεταφέρουν και θα την εφαρμόσουν στη συνεχεία. Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα θα έλεγα ποτέ δεν συμβαίνει αυτό με βάση τη μελέτη μας. Δεύτερον, η άλλη σύσταση είναι να εξασφαλίσουμε ότι όταν είναι όταν υπάρχει θέμα χρόνου ε, για την εφαρμογή, τότε θα πρέπει, για να μεταφερθεί δηλαδή η σχετική νομοθεσία, τότε να χρησιμοποιούμε καλύτερα κανονισμό παρά οδηγία. Εδώ το Κοινοβούλιο μπορεί να πιέσει την Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι η παρακολούθηση και η εφαρμογή της οδηγίας των κανονισμών, των, ε, συγγνώμη, και η εφαρμογή των κανονισμών γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι οδηγίε. Γιατί συνήθω δεν γίνονται με τον ίδιο συστηματικό τρόπο. Και αν κοιτάξουμε στην ετήσια, ε, σε αιτήσει εκθέσει, βλέπουμε ότι έχουμε διαφορετικού τύπου πληροφορίε για τα μεν και τα δε. Τώρα, όταν μιλάμε για τα διάφορα εργαλεία προώθηση τη συμμόρφωση που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να προωθήσει την εφαρμογή. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει πιο στρατηγική προσέγγιση στη χρήση αυτών των εργαλείων. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Κάποια από αυτά τα μέσα, θα πρέπει, οι συστάσει θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο συστηματικά και κάποια άλλα μόνο όταν υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένες ανάγκες τη οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί. Μπορείτε να κοιτάξετε την ανάλυση των διαφόρων εργαλείων. Θα ήθελα να σας τονίσω όμως ότι οι μελέτες που ελέγχουν τη συμμόρφωση και την ε, μεταφορά ε, του ενωσιακού δικαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, συστηματικά, καθώς και τα σχέδια μεταφοράς και εφαρμογής, καθώς και όλα τα μέσα που προβλέπει η διαδικασία επί Για την υποχρεωτική χρήση των πινάκων συσχετισμού, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατά επανάληψη στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να τα χρησιμοποιήσει αυτά, να τους χρησιμοποιήσει. Και νομίζω ότι αυτό το, και αυτό το Κοινοβουλίο θα πρέπει να προωθήσει αυτό το θέμα. Υπάρχουν δύο διαθεσμικέ ε, συμφωνίε μεταξύ του, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη δίνουν τέτοιου πίνακε ε, ε, συσχετισμού για την ε, μεταφορά των νομοθετημάτων. Και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι η Κομισιόν το κάνει και ότι έχει επαρκή πόρου για να το εξασφαλίσει. Γιατί είναι ο μόνο τρόπο για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει σωστή εφαρμογή τη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου. Επιπλέον, υπάρχουν και οι επιθεωρήσεις ε, σε ενωσιακό επίπεδο από ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς. Αυτό το έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορες φάσεις τα τελευταία χρόνια θεωρείται απαραίτητο να γίνονται τέτοιες επιθεωρήσεις ή έρευνες αν θέλετε για τις περιπτώσεις ή ε, παράπονα ε, παραβάσεων στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτής της αρμοδιότητας, αυτές τις εξουσίες. Και όταν τίθεται στο δικαστήριο ένα συγκεκριμένο θέμα, δεν έχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξουν μια υπόθεση και μερικέ φορέ χάνουν την υπόθεση, χάνουν υπόθεση κομισιών. Έχουμε παραδείγματα όπου γίνονται επιθεωρήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. για την ευημερία των ζώων, για τα θαλάσσια θέματα, για την ασφάλεια των τροφίμων και δεν υπάρχει κανένα λόγος για το περιβάλλον, που είναι αρκετά περίπλοκο θέμα, να μην έχουμε αντίστοιχε επιθεωρήσεις που θα συμπληρώσουν απλώ. το μηχανισμό follow-up των ε, διαδικασιών ε, παραβάση και των πιλωτικών διαδικασιών της Κομισιόν. Σε σχέση με, την, ε, με το enforcement, την εφαρμογή, υπάρχουν δύο βασικά εργαλεία, τα πιλωτικά και οι διαδικασίες επιπαραβάση. Τα πιλωτικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η φάση που γίνεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση και είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε το 2007 με πρωτοβουλία της Κομισιόν δεν έχει την δική του νομική βάση αυτό το εργαλείο στην συνθήκη και σκοπό έχει να διορθώσει προβλήματα συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο, δημιουργώντας πλατφόρμες που, συνδέει, που συνδέουν την Κομισιόν με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Ο άλλος στόχος είναι να, μειωθεί, να μειωθούν βεβαίως οι παραβάσεις και τρίτος, να προσπαθήσει να δώσει πιο γρήγορες απαντήσεις στους πολίτες και στα παράπονα των πολιτών. Τα πρόβλημα με το πιλωτικό αυτό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έλλειψη νομικής βάσης. Εάν λάβουμε υπόψη τη διαδικασία επιπαραβάση, άρθρο 258, το άρθρο αυτό δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα τη στιγμή που τα κράτη-μέλη έχουν παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις. Καταρχήν αποστέλλεται επίσημη επιστολή στα κράτη-μέλη. By the The... και υποβάλλεται στη συνέχεια αιτιολογημένη γνώμη. Άρα, μέσα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι η θέση των κρατών μελών και τις παρατηρήσεις τους, αλλά δεν υπάρχει νομική βάση. Ε, ως προς αυτό τον κλειστό διάλογο μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαδικασία αυτή αμφισβητήθηκε για δύο λόγους. Αρκετές φορές Ο διάλογος αυτός είναι σχηνοτενής, ε, διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, ε, δηλαδή υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της διαδικασίας αυτής. Άρα πρόκειται για μία μακρά περίοδο μη συμμόρφωσης των κρατών μελών. Άρα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς, διότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, συμμορφώνονται, ενώ άλλα έχουν την δυνατότητα μη συμμόρφωσης για μία μακρύτερη χρονική περίοδο. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το EU Pilot αμφισβητείται είναι ότι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, διότι αυτές ε, οι αποφάσεις ε, λαμβάνονται σε ε, καθαρά περιορισμένο επίπεδο και στη συγκεκριμένη περίπτωση και από ό,τι βλέπουμε από τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου μελέτησαν περισσότερες από 2.800 πρόσφυγες. Οι 621 οδήγησαν σε EU Pilot. Οι υπόλοιπε δεν εκδικάστηκαν καν. Πρόκειται δηλαδή για πολύ υψηλό αριθμό. Στις συστάσεις μας λοιπόν αναφέρουμε ότι χρειάζεται έλεγχος νομιμότητας μέσα στην όλη διαδικασία. Εγκρίνοντας κανόνες όπου ορίζουμε το χρονικό διάστημα της κάθε διαδικασίας καθώς και το ρόλο των διαδίκων. Η διαδικασία επί αναγνωρίζεται ευραίος. δηλαδή από τη στιγμή της παράβασης το κράτος μέλος γνωρίζει ότι το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στο, στο δικαστήριο. Με συγχωρείτε. Άρα ε, αυτό το βήμα είναι πολύ σοβαρό. Η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει τη χρήση αυτής της διαδικασίας. Άρα στις συστάσεις μας ορίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός που να ορίζει τους κανόνες για το EU Pilot αλλά και για τη διαδικασία επιπαραβάση για να δούμε πώς θα οριστεί το κάθε βήμα και πότε αρχίζει ένα EU Pilot, πότε λύγει και Οπότε ξεκινά η διαδικασία επί παραβάση. Υπάρχει ένα θέμα και ε, νομιμότητας του EU Pilot, διότι οι ε, εναγόμενοι δεν συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Όπως και στη διαδικασία επί παραβάση. Η συμμετοχή του ενάγοντα μπορεί να οδηγήσει σε ακριβείς πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα την επιχειρηματολογία της Επιτροπής και των κρατών μελών. Άρα, η διαδικασία παράβασης οδήγησε σε ταχεία επίλυση των υποθέσεων. Αυτό το είδαμε στην Ιταλία ιδιαίτερα και θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, εναγόντων αλλά και του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να λάβει πληροφορίες από τις προσφυγές που αποστέλλονται στην Επιτροπή και να συμμετέχει στη διαδικασία μέσα στα πλαίσια του EU Pilot ή εποπτεύοντας αυτή τη διαδικασία. Και το τελευταίο θέμα είναι η διαφάνεια της διαδικασίας επί παραβάση. Το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να δώσει στοιχεία μέσω μιας τράπεζης δεδομένων ως προς τη διαδικασία επιπαραβάση, ποια κράτη-μέλη αφορά και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή η τράπεζα δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι απαρχαιωμένη και δεν δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι ρόλος του Κοινοβουλίου σε αυτή τη θητεία είναι να ζητήσει από την Επιτροπή να ενημερώσει αυτή την βάση δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία μου για αυτή την πολύ σημαντική εισήγηση. Και τώρα έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για τις άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τους ε, δύο πρώτους ομιλητές, Χόιζελ και Στότς. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή υπάρχει ε, έλλειψη αποτελεσματικότητας ή ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων ή του ε, κάθε ποινικού συστήματος, διότι υπάρχει μία γκρίζα ζώνη όταν ε, και εκεί που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο. Δηλαδή ένα κράτος μέλος θα πρέπει να εμπιστεύεται το δικαστικό σύστημα ενός άλλου κράτους μέλους το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, διαδραματίζει κάποια, κάποιο ρόλο. Κυρία Μπαλεστέρος, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να δώσουμε επίσημο χαρακτήρα στο EU Pilot και να ξαναδούμε τις διαδικασίες επί παραβάση. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας υποβάλω πολύ συχνά ομάδες της κοινωνίας των πολιτών ε, εμπιστεύονται τη, τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, θεωρούμε ότι πρόκειται για ε, θεμα, μεγάλο θεματοφύλακα των συνθήκων. Εδώ μιλώ για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πιστεύω ότι πολλές φορές τα αποτελέσματα της Κομισιόν είναι άκρος απογοητευτικά. γιατί πολλές φορές ε, στεκόμαστε σε οικονομικά συμφέροντα και όχι στην προστασία. Δηλαδή στερούμε στα περιβαλλοντικά ως προς τον ε, κανονισμό για τις ευθύνες έναντι του περιβάλλοντος. Μπορείτε να μας πείτε πώς εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Ίσως θα πρέπει να δούμε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτή η οδηγία. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις, δύο ακόμα μιλητές. Θα ομοδοποιήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε στις απαντήσεις. Ο κύριος Πίντου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες σκέψεις πριν Υποβάλλω ερωτήσεις προς τους τρεις ομιλητές. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση έναντι του κοινοτικού δικαίου, το οποίο είχαμε παραμελήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λαμβάνουμε υπόψη την κοινοτική ένωμη τάξη η οποία τάσεται υπέρ του εμπορίου, των συναλλαγών και των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μετασχηματισμό της ΕΟΚ, που ήταν μετεξέλιξη της ΕΚΑΧ. Πρόκειται λοιπόν μία μερκαντιλιστική προσέγγιση του θέματος. Ήδη από την πρώτη αυτή απαρχή του δικαίου, κύριο μας μέλημα είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα. Απαρτιζόμαστε από 28 κράτη-μέλη, δηλαδή 28 ένομες τάξεις που διαφέρουν. Αυτό ίσως φαίνεται πρόβλημα, αλλά ίσως και να μην είναι. Το δίκαιο διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες αρχές. Οι νόμοι δεν είναι το δίκαιο. Δίκαιο είναι και η νομολογία και το εθιμικό δίκαιο. Το κράτος δικαίου βασίζεται στο δίκαιο. Και τι σημαίνει δίκαιο. Εθνικά δικαστήρια. Υπάρχει ένα δικαιοδοτικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το κύριό μας ε, μέλημα δεν είναι ο άνθρωπος και υστερούμε και στο ποινικό. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη είναι ότι εμείς δεν θεωρούμε τον άνθρωπο παρά εγκληματία. Μιλάμε για τρομοκράτες, εγκληματίες, αλλά εδώ θα πρέπει να θέσουμε την γραμμή οριοθέτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα αυτά. Η διάρθρωση του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα ως προς το ποινικό, αφορά την κατάρτιση ορισμένων βασικών νόμων που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Το τεκμήριο της ε, αθωότητας, για παράδειγμα. Κανένας δεν μπορεί να καταδικαστεί χωρίς να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υπάρχει και το δικαίωμα στην προσφυγή και το δικαίωμα στην υπεράσπιση. Θα ήθελα να σταθώ σε μία ιστορία που όλοι γνωρίζουμε αλλά ίσως δεν είναι γνωστή με αυτή τη διάσταση. Πριν από χιλιάδες χρόνια δικάστηκε κάποιος στη Γαλιλαία. Την πέμπτη το βράδυ καταδικάστηκε και στη συνέχεια σταυρώθηκε. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια επιτάχυνση του δικαιοδοτικού συστήματος που στην ουσία αφαιρούν το δικαίωμα στην υπεράσπιση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν τον ε, Ναζωρέο, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος ε, καταδικάστηκε. Όμως, εγώ διάλεξα να είμαι δικαστής και δικηγόρος, διότι θεωρώ ότι ο υπόδικος έχει δικαίωμα στην ε, υπεράσπισή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είχαν και ήταν, είχαν υπερασπιστεί αυτό τον άνθρωπο, στην ουσία σιώπησαν την ώρα της δίκης. Οι δικηγόροι είναι η πεμπτουσία του δικαίου και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον ε, πολίτη και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανεξαρτησία του δικαιοδοτικού συστήματος και του δικαστή. Το ερώτημα λοιπόν τώρα που θέλω να υποβάλω στους τρεις ομιλητές είναι το εξής. Μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπόδια έτσι ώστε να γίνει τυποποίηση όλων των βαθμών αδικημάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση και σε αυτό τον τομέα, διότι ό,τι είναι ποινικό σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να έχουμε μία ένομη τάξη σε έναν μόνο τομέα. Θα πρέπει να διαθέτουμε ένομη τάξη σε όλους τους τομείς. Έτσι ώστε να υπάρξει και ένα κοινό ποινικό σύστημα, ε, δημιουργώντας μία τυποποίηση. Να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή έτσι ώστε ε, να λάβουμε υπόψη όλα τα αδικήματα. Το αδίκημα της εξαπάτησης, το, την, ε, περίπτωση της δυσφήμισης, όλα τα στάδια και όλους, όλες τις βαθμίδες των αδικημάτων που θα πρέπει να πλαισιώνονται από ένα ενιαίο, ε, μια ενιαία ένομη τάξη. From Άλλη μια ερώτηση θα ακούσουμε από την κυρία Μορβάη και μετά πρέπει βεβαίως να ακούσουμε όχι μόνο τις ερωτήσεις αλλά να έχουμε και χρόνο για απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ωραίο είναι όταν ε, ο νόμος και το πάθος ε, πάνε χέρι με χέρι. Η δική μου ερώτηση θα είναι πολύ πιο βαρετή. Αφορά τις ε, παρεξηγήσεις για την εφαρμογή της ε, χάρτας ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφέρατε, ανάφεραν δύο μιλητές περιπτώσεις οποίες δεν είχε εφαρμογή η χάρτα Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόστηκε στα εθνικά δικαστήρια η χάρτα. Ε, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλάω και να μιλάει και ο διπλανό, η διπλανή μου συνέχεια σε άλλη γλώσσα. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη. Αν μπορείτε λίγο να με ακούσετε. Ευχαριστώ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι νομολογία υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εφαρμογή της χάρτας, είτε μιλάμε για εθνικά δικαστήρια, είτε για το 10. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Δεδομένου του ότι η κυρία Μορβάη ήταν τόσο σύντομη, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και τον κύριο Μπρετόν με την τέταρτη ερώτησή του. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σε πιστήσω την προσοχή αγαπητοί ομιλητέ, σε δύο προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν εντάχει. Καταρχά, την αρχή τη υπεροχή, που είναι μια αρχή του δικαίου που δημιουργήθηκε το 1964 από την απόφαση Κώστα. Είναι σημαντική αυτή η απόφαση γιατί η νομολογία λέει ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει υπεροχή ακόμα και έναντι των συνταγμάτων των κρατών μελών. Και εδώ υπάρχει ένα δημοκρατικό σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, για ένα... Είναι τόσο σημαντική αυτή η αρχή και όμως δεν υπάρχει πουθενά στην συνθήκη. Υπήρχε στο σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος, ξεκάθαρα, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι εγκαταλείφθηκε μετά από το αρνητικό δημοψήφισμα, ειδικά του γαλλικού λαού, και η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ενσωμάτωσε ένα μεγάλο τμήμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, δεν μιλάει για αυτή την αρχή της υπεροχής. Επομένως, το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, δεν είναι προβληματικό το ότι δράζουμε το σύνολο του ευρωπαϊκού δικαίου πάνω σε μία αρχή που δεν μπορέσαμε να την εσωματώσουμε στην συνθήκη που επικύρωσαν τελικά τα κράτη-μέλη. Είναι δεύτερον φυσιολογικό ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να δημιουργεί μια τέτοια τόσο σημαντική αρχή που ανατρέπει πολλά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο τώρα. Όλοι χαίρονται που ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων υιοθετήθηκε και μερικοί λυπούνται που δεν εφαρμόζεται επαρκώς ακόμα και σήμερα. Ένα πρόβλημα που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διασφάλισης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 1950 και από τη μία και από την άλλη χάρτα. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, διατυπώνται με παρόμοιο τρόπο στα δύο κείμενα και τα δύο κείμενα τα προστατεύουν διαφορετικά δικαστήρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, προστατεύει τη σύμβαση του 1950 και το, το άλλο προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπορεί να υπάρξει ε, σύγκρουση εδώ πέρα. Ε, δεν θα θέλαμε να υπάρχουν τέτοιου τύπου συγκρούσει ανάμεσα σε τέτοιου τύπου κείμενα. Thank you very much, and Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Με τη σειρά που επιθυμείτε. Σε δύο λεπτά όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με τη σειρά που μιλήσατε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης δεν αμφισβητείται, το δείχνουν και τα νούμερα της Κομισιόν. Ο χρόνος έκδοσης έχει μειωθεί τόσο πολύ, ώστε μιλάμε για επιτυχία. Εγώ δεν έχω ακούσει ε, διαδικασίες σε παραβάση για την ανεξαρτησία των δικαστηρίων που αποφασίζουν για αυτές τις υποθέσεις, αλλά βεβαίως ε, η κατασκευή έχει αναγκάζει τα δικαστήρια να εκδώσουν ένα ένταλμα σύλληψης εάν συντρέχουν ε, όλες οι προϋποθέσεις. Δεν τίθεται ζήτημα διακριτικής ευχέρειας αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν επιθυμητό και είναι λογικό σε μια κοινότητα δικαίου που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το εάν δικαιολογείται αυτή είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό μπορεί να ισχύει και στο εσωτερικό μιας χώρας. Εάν υπάρχει τώρα ζήτημα παραβίασης ανθρωπίνων ή θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι πλέον ζήτημα του ΔΕΚ σε ε, τέλεση βαθμό να κρίνει γιατί βεβαίως πρόκειται για εφαρμογή ενός μέσου του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, επί της αρχής, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην πράξη βεβαίως μπορεί να υπάρχει. Το πραγματικό πρόβλημα είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις ε, χρησιμοποιείται με τρόπο όχι πολύ αναλογικό. Και θα ήθελα να πω στον κύριο Μαρίνιου Πίντου πως ε, εκτιμώ το ότι ζητήσατε περισσότερη ενότητα στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, αλλά πρέπει να περιοριστεί νομίζω όπως λένε και οι συνθήκες σε αυτά τα οποία ισχύουν ε, διασυνοριακά και μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση του ποινικού δικαίου μόνο σε τομείς που υπάρχει αυτό το διασυνοριακό στοιχείο. Οπότε υπάρχει ακριβώς ε, και αυτό το οποίο λέμε ενωμένη στην ε, πολυμορφία. Αν τα κριτήρια της ληστείας ή της δολοφονίας είναι διαφορετικά, ε, ας είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα σχέση με το άλλο ερώτημα, υπήρχαν αρκετά για τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα αφήσω την, την απάντηση αυτή στον κύριο Στότς. Ε, για τον κύριο Μπρετόν βεβαίως και για το πιο δίκαιο κατησχεί πράγματι ε, μπορούμε να συζητάμε δύο μέρες. Κοιτάξτε, βεβαίως στην αρχή ήταν δικαστική η εξέλιξη, όλα τα κράτη-μέλη σε όλες τις επόμενες αναθεωρήσεις της συνθήκης αναγνώρισαν το κεκτημένο ως έχει και άρα και την ομολογία του ΔΕΚ, άρα θεωρώ εγώ και την ερμηνεία αυτή. Βεβαίω πάντα υπό την επιφύλαξη των ε, συνταγματικών δικαστηρίων, ειδικά της χώρας μου από πλευρά συνταγματικού δικαίου, αλλά και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε σε συναρπαστικές διασκέψει κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις ήταν βεβαίως πολιτικής φύσης, βεβαίως το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο ε, αναγνωρίζει αυτά τα οποία γράφονται στις οδηγίες για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κτλ. δεν τίθεται ζήτημα. Ε, δεν ασκεί πολιτική, απλά ερμηνεύει τους νόμους μόνο το δικαστήριο. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αυτό το ερώτημα να απευθύνεται στο Κοινοβούλιο. Το πώς διαμορφώνονται δηλαδή οι οδηγίες, ε, μέχρι πού πηγαίνει η αναγνώριση διαφορετικών ενιών του δικαίου. Αυτό είναι ζήτημα περισσότερο πολιτικής ε, του δικαίου. Τώρα, το τρίτο ερώτημα για την εφαρμογή της χάρτας. Βεβαίως, ε, το δικαστήριο χρησιμοποίησε τη χάρτα σε πολλές περιπτώσεις και στις περισσότερες από αυτές τα ερωτήματα ήταν από εθνικά δικαστήρια. Να σας υπενθυμίσω το δικαστήριο συχνά ε, κατηγορείται πως καθυστερούσε πριν ε, υπάρξει η, κάρτα, η χάρτα αυτή όσον αφορά την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό πλέον δεν ισχύει εφόσον είναι εν ισχύ η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο την εφαρμόζει και σε διοικητικές αλλά και σε ε, περιπτώσεις ε, νομοθετικές. Είχαμε δηλαδή νομοθετήματα του Συμβουλίου, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τα οποία ε, καταρρίφθηκαν γιατί θεωρείται πως δεν είναι συμβατά με τελευταίο και τρανό παράδειγμα βεβαίως την νομοθεσία για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, η οποία αντιβαίνει στο άρθρο 7, το λεγόμενο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κτλ. Έχουμε λοιπόν από το δικαστήριο ένα πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο του κατά πόσον το δευτερογενές δίκαιο συμμορφώνεται με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και μπορώ να πω πως εμπνέεται το δικαστήριο και θέλει να εφαρμόσει την Χάρτα αυτή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μπορώ να σας ε, στείλω έναν κατάλογο αν θέλετε, στον οποίο ε, πράγματι εφάρμοσε το δικαστήριο τα όσα αναγράφει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τελευταίο ερώτημα, ποιο, αν κατησχύει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Εθνικού και από πλευράς ε, συνταγματικής. Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συνεχώς. Και από την εμπειρία μου σπάνια προκύπτει ζήτημα. Εγώ μία περίπτωση γνωρίζω όπου πράγματι το δικαστήριο είπε πως συνταγματική διάταξη κράτους μέλους ε, είναι ε, αντίθετη με τη συνθήκη και ήταν νομίζω πριν από 20 χρόνια όταν αποφάσισε το δικαστήριο πως η απαγόρευση που υπήρχε στο γερμανικό σύνταγμα ότι οι γυναίκες ε, δεν επιτρέπεται να έχουν μάχημες θέσεις ε, στο στρατό ε, αντιβαίνει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αλλά νομίζω ήταν θετική η υποδοχή στη Γερμανία. Υπήρξε συνταγματική αλλαγή και σήμερα υπηρετούν οι γυναίκες στο στρατό της Γερμανίας. Θεωρητικά δηλαδή υπάρχει το πρόβλημα, αλλά... Αλλά δεν μιλάμε και για ανατροπή. Είναι μια λογική αρχή αυτή θα έλεγα. Αναφέρεται και στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας και κατά την άποψή μου είναι μια αναγκαία αρχή. Και δεν πρέπει να τη βλέπουμε ξεκομμένη αλλά σε συνδυασμό με άλλες ε, διατάξεις της ε, συνθήκης. Επίσης η συνθήκη σε ένα από τα πρώτα άρθρα εγγυάται το δικαίωμα στην εθνική ταυτότητα. Έτσι, οπότε το ότι η του εθνικού δικαίου ε, σε, πρέπει να το δούμε σε αντιδιαστολή με το δικαίωμα στην εθνική ταυτότητα. Έτσι. Και νομίζω το ένα αντισταθμίζει το άλλο. Το άλλο ερώτημα ήταν... Η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ Εστρασβούρου και Λουξεμβούρου. Στο άρθρο 6 της συνθήκης αναφέρεται ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γίνεται μέλος ε, της ε, προσχωρή στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το ξέρετε, όπως και εγώ, διαπραγματεύτηκε την ένταξή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα κείμενο της σχετικής σύμβασης και εκεί πέρα ρυθμίζεται το ότι το δικαστήριο του Στρασβούργου θα μπορεί να κρίνει και περιπτώσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το κείμενο αυτής της συμφωνίας αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι στο δικαστήριο γιατί ζήτησε μια αιτιολογημένη γνώμη ή η Κομισιόν η συζήτηση έγινε και υποθέτω πως ε, η απόφαση θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες. Οπότε επί της ΟΣΕΑΣ, επειδή είναι μια υπόθεση η οποία εκρεμεί ακόμα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά μπορώ να σας πω πως ε, υπάρχει μια ανταλλαγή και επαφή των δικαστών Λουξεμβούργου και Στρασβούργου συναντώνται τακτικά και ε, το δικαστήριο του Λουξεμβούργου επίσης έχει τακτικές συναντήσεις με τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών ειδικά τα συνταγματικά δικαστήρια. Υπάρχουν και ανταλλαγές μεταξύ του Γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και του ΔΕΚ στο Λουξεμβούργο. Και Αυτά δεν είναι απλές ε, έτσι, τυπικές συναντήσεις για να γίνουν χειραψίες, αλλά είναι διασκέψεις ε, που εξετάζουν την συνεργασία, την ερμηνεία, είναι πάντα πάρα πολύ επικοδομητικές ε, ανταλλαγές απόψεων και εκεί πέρα νομίζω ακριβώ πως περιορίζεται ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης. Θεωρητικά δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά νομίζω πως δεν είναι πολύ σοβαρή πιθανότητα. Ευχαριστώ. Um, Θα περιστώ σε απαντήσεις, σε ερωτήσεις για την περιβαλλοντική ευθύνη και τις ερωτήσεις του κύριου Μαρινό Κάμπους. Έχουμε δύο οδηγίες για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν περιβαλλοντικές οδηγίες και σκοπό έχουν να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον. Δεν υπάρχουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα αντιδράσουν ε, για να εξασφαλίσουν την προστασία της. Οι μηχανισμοί εφαρμογής που υπάρχουν ε, μέσω της διαδικασία παραβάσης και των, ε, περιβαλλοντικών, και των πιλωτικών σχεδίων είναι πολύ σημαντικά για αυτές τις οδηγίες. Και οι αποτυχίες, η έλλειψη διαφάνειας, η καθυστέρηση της Κομισιόν για να αντιμετωπίσει κάποια αυτά τα θέματα ή τα προβλήματα παράβασης αυτών των δύο οδηγιών είναι πιο σημαντικά σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι οδηγίες είναι εύκολο να τις παρακολουθήσει κανείς, δηλαδή οι πολίτες να τις παρακολουθήσουν. Οι πολίτες μπορούν να δουν πότε κάποια είδη, ας πούμε, του ζωικού κεφαλαίου κτλ. Ε, εξαφανίζονται. Ενώ μπορεί να υπάρχουν άλλες οδηγίες περιβαλλοντικέ που είναι πιο τεχνικές και οι πολίτε δεν μπορούν να συλλάβουν τα προβλήματα. Δεν είναι Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι συστάσει που έχουμε προτείνει για να καταστούν πιο αποτελεσματικά αυτά τα μέσα που έχουμε ε, στα πλαίσια των πιλωτικών σχεδίων και των διαδικασιών οι επιπαραβάσεις είναι πολύ σημαντικά, ειδικά για την οδηγία, για, την, για τα οικοσυστήματα και για την η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Εδώ η Κομισιόν θέλει να υιοθετήσει μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Κάναμε μια μελέτη για τον λογαριασμό της Κομισιόν για την εφαρμογή και για την ευθύνη για ζημίες, έχουμε δει ότι υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης για την κατανόηση αυτής της οδηγίας και της οδηγίας για τα οικοσυστήματα και έλλειψη εναρμόνισης για την κατα... από της κατανόησης όλων των κρατών μελών, όπου κράτη-μέλη, πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτή η οδηγία αφορά τις περιπτώσεις όπου έχουμε ζημιές που προσεδιάζουν σε καταστροφές, τρομακτικές ζημιές δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι στις άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν απλώς ε, ζημιές στην βιοπικιλότητα, αυτός που πληρώνει είναι το κοινό. Δηλαδή οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να βρουν τις λύσεις στις ε, ζημιές που έγιναν ε, στη βιοπικιλότητα και όχι στους, σε επιχειρήσεις ας που δημιούργησαν το πρόβλημα. Εάν εφαρμοστούν όμως αυτές οι οδηγίες και αν εφαρμοστούν για όλες τις ζημιές και όχι μόνο για αυτές τις τρομακτικές ζημιές που μοιάζουν με καταστροφή, τότε οι υπεύθυνοι φορείς, ε, εταιρείε κτλ. θα πληρώσουν για αυτές τις ζημιές. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε αυτή τη φάση. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η Κομισιόν με την επόμενη έκθεση που θα ετοιμάσει το 2014. Και ελπίζω να υπάρξει και σωστή αναδιατύπωση ε, της οδηγίας μετά από τη συνειδητοποίηση αυτή. Ευχαριστώ. Σύντομα μάλιστα. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές για τις απαντήσεις. Στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών προχωρούμε τώρα στο δεύτερο μισό της ακροασής μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον, στην καθηγητή Ξάντρα Κράμερ που θα μας ταξιδέψει λίγο σε ένα θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ο τίτλο της παρέμβασή τη. Έχετε το λόγο. Σα um, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σταθώ στο ιδιωτικό διεθνές ε, δίκαιο και όπως ξέρετε νοείται ότι καλύπτει θέματα διεθνούς ε, δικαιοδοσίας και τι ισχύει στις ε, διασυνοριακές σχέσεις και την εφαρμογή, την ισχύ ε, ενός ε, διεθνούς νόμου. Δυνάμει του άρθρου 81 για τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ένα επιπρόσθετο κομμάτι το οποίο θα με απασχολήσει μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, διασυνοριακής ε, αντιμετώπισης του ιδιωτικού δικαίου. Με απασχολεί λοιπόν το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο μέσα στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου με βάση το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο που μας διέπει τα τελευταία 15 χρόνια. Επίσης, στάθηκα και στο νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα καθώς και τις μελέτες που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου συμμετείχα και εγώ. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σταθώ εν συντομία σε όλους αυτούς τους τομείς και αν θέλετε μπορείτε να δείτε και το γραπτό μου κείμενο για περαιτέρω πληροφορίες επί των θεμάτων. Βεβαίως στον στομέα, το στομέα του αστικού δικαίου, δυνάμει του άρθρου 81, μιλάμε για τις ελευθερίες, ασφάλεια και τη δικαιοσύνη και βλέπουμε ότι το ιδιωτικό δίκαιο αποτελεί την πεμπτουσία της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς διότι διευκολύνονται οι διασυνοριακές σχέσεις για τα φυσικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Τα μέσα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αφορούν την ασφάλεια των σύναλλων αρχών την κατανομή δικαιοδοσίας μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση διαφοράς και τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη-μέλη. 15 χρόνια πριν, η συνθήκη δημιούργησε ε, ειδικές σχέσεις και μία παρέκταση σχέσεων και σε εμπορικά ζητήματα δυνάμει του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Υπάρχει όμως ένας περιορισμός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αφορά το οικογενειακό δίκαιο, διότι το άρθρο 81 προαπαιτεί ομοφωνία σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό ε, το οικογενειακό ε, δίκαιο μπορεί να ισχύσει διασυνοριακά με βάση την ομοφωνία. Και αυτό έθεσε ορισμένα προσκόμματα στο παρελθόν, δηλαδή την εφαρμογή του κανονισμού ΡΟΜ 3. Δεν ήταν δυνατόν να φτάσουμε σε ομοφωνία και γι' αυτό αυτός ο κανονισμός εγκρίθηκε με βάση την ενισχυμένη συνεργασία. Επίσης υπάρχουν προτάσεις που εκκρεμούν θα ήθελα να αναφερθώ στις καταγεγραμμένες εταιρικές σχέσεις που υπάρχει, όπου υπάρχει διαφορά σε σχέση, υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου. Και εάν δούμε το γενικότερο πλαίσιο, μπορούμε να δούμε ότι οι περιορισμοί αυτοί του οικογενειακού δικαίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη Εάν δούμε την πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία 15 χρόνια, έχει υποστηρίξει το νομοθετικό ε, πλαίσιο και βλέπουμε ότι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να οικοδομήσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι ότι βεβαίως υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και γι' αυτό υπάρχει και η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων. Θα πρέπει όμως να οικοδομήσουμε αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γι' αυτό αυτή η οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασίζεται στο ρόλο των κρατών μελών. Δέκα χρόνια πριν αναγνωρίσαμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο συνεκτικός ε, κρίκος, αυτή η συνοχή, γιατί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε παρά με ορισμένους τομείς. Και βλέπουμε ότι μεταξύ αυτών των ε, μέσων υπάρχει έλλειψη συνοχής. Άρα πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε ένα σαφές δικαιοδοτικό πλαίσιο. Πρόσφατα επίσης έχουμε σταθεί στην οικονομική ανάπτυξη, στην κινητικότητα των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων ιδιαίτερα προς τον κανονισμό περί αφαιρεγγιότητας. Εδώ γίνεται λόγος για αναδιάρθρωση επιχειρήσεων για να εξασφαλίσουμε την οικονομική τους ανάκαμψη. Εάν δούμε τα έγγραφα γενικότερων πολιτικών ή πολιτικής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου, καθώς και την ατζέντα της Κομισιόν για το 2020, Μιλάμε για ε, εδραίωση, ε, παγίωση και ενιαία εφαρμογή. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι εργασίες του 2000 που άρχισαν το 2012 από το ε, Κοινοβούλιο αφορούν ένα πιο συνεκτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Αν δούμε λοιπόν τι έχει γίνει μέχρι τώρα δυνάμει του άρθρου 81% στη δικαστική συνεργασία σε αστικά ζητήματα βλέπουμε ότι σε 15 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. 13 ε, κανονισμοί ασχολούνται με την πεμπτουσία του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και για την αμοιβαία αναγνώριση και εφαρμογή. Ενώ παράλληλα υπάρχει σωρία κανονισμών που ασχολούνται ασχολούνται με υπολοιματικά ζητήματα σε σχέση με την τεκμηρίωση και τα αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης υπάρχουν και δύο ε, οδηγίες που αφορούν τη δικαστική αρρωγή ε, η οποία ορίζεται διασυνοριακά. Υπάρχουν ε, τρεις προτάσεις που εκκρεμούν. Επίσης υπάρχουν οδηγίες που έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 114 της Συνθήκης στα πλαίσια της γενικής εναρμόνισης που σχετίζονται με την ε, δικαστική συνεργασία. Έχουμε να κάνουμε και με περιπτώσεις ε, διασυνοριακών υποθέσεων. Εδώ βλέπουμε διάφορους ε, κανόνες που ισχύουν ανάλογα με το που βασιζόμαστε στη συνθήκη. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ερμήνευσε τα διάφορα μέσα και προσέθεσε στο γενικό αυτό πλαίσιο, δηλαδή η νομολογία που αφορά την ελεύθερη εγκατάσταση επιχειρήσεων έχει βοηθήσει ιδιαίτερα, καθώς και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, οι αποφάσεις περί ευρωπαϊκής ηθαγένειας που έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα στην εφαρμογή ιδιωτικού, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. και βεβαίως και η ελεύθερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων που βοήθησε και στην εφαρμογή του εταιρικού δικαίου. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη συνθήκη της Χάγης για την εφαρμογή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Πολλά κράτη-μέλη έχουν εγκρίνει τη συνθήκη και καθίσταται σαφές ότι στο μέλλον αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχόλησε μέσα στα πλαίσια μιας μελέτης είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ε, ενδοκινοτικών μέσων και τρίτων χωρών. Τα περισσότερα μέσα ή μηχανισμοί που διαθέτουμε περιορίζονται στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά οι διασυνοριακές σχέσεις δεν σταματούν στα κοινοτικά σύνορα. Γι' αυτό ασχολούμαστε και με πολίτες από τρίτες χώρες που ζουν στα κράτη-μέλη, ζουν και εργάζονται. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διενεργηθεί μία μελέτη για τα χάσματα που υπάρχουν μέσα ε, στα πλαίσια των εργασιών, καθώς και την εφαρμογή ενός πιο ε, συνεκτικού πλαισίου που να διέπει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Είπαμε λοιπόν ότι στα πλαίσια του μη οικογενειακού δικαίου και στα πλαίσια του εταιρικού δικαίου, επειδή υπάρχουν ε, σοβαρά χάσματα και δεν υπάρχει κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα καλύψουμε. Επίσης, θα πρέπει να δούμε να σταθούμε με το δικαίωμα για τον ιδιωτικό βίο με βάση και την εφαρμογή του κανονισμού Ρόμ 2. Το Κοινοβούλιο ψήφισε το 2012 επί του θέματος, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί συνέχεια ως προς την προσφυγή, συλλογική προσφυγή σε ένδικα μέσα. Υπάρχει μια σύσταση της Επιτροπής επί του θέματος, θεωρούμε όμως ότι χρειάζεται μία πιο εκτενής προσέγγιση του θέματος της προσφυγής στα ένδικα μέσα με βάση το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Στο οικογενειακό δίκαιο υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα χάσματα διότι έχουμε νομοθετήσει πολύ πιο πρόσφατα και το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο γιατί προαπαιτείται ομοφωνία για να εγκριθούν, τα, να εγκριθούν μέσα που να διέπουν το οικογενειακό δίκαιο. Και επίσης το ουσιώδες ε, δίκαιο θα πρέπει να διέπεται από γενικές αρχές που διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ όλων των μέσων και υπάρχει και ένα είδος ε, διά, ε, διάδρασης όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο ή άλλες ε, πτυχές του εμπορικού δικαίου. Και αυτό αφορά και το δικαίωμα της εγκατάστασης όπου βλέπουμε ασυνέπειες τα ad hoc μέσα οδήγησαν σε επαναλαμβανόμενους ε, κανόνες εφαρμογής. Πολλές φορές όμως ε, αλλάζει το πλαίσιο και η ουσία. Αυτό που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, μία μελέτη κόστους ωφελίας, να δούμε δηλαδή ότι το συνολικό κόστος είναι της τάξης του, των 140 εκατομμυρίων ετησίως για να καλύψουμε αυτό το, το πλαίσιο ασυνέπειας. Τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ε, αν σταθούμε στον ελάχιστο παρονομαστή, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το ε, πλαίσιο που μας διέπει και να σταθούμε, να προχωρήσουμε μάλλον και στο μη οικογενειακό δίκαιο, γιατί εκεί δεν χρειάζεται, δεν προαπαιτείται ομοφωνία. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με το εταιρικό δίκαιο. Όπως γνωρίζετε, λίγους μήνες πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να διενεργηθεί η μελέτη για το εταιρικό δίκαιο και πώς εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις και είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει το Κοινοβούλιο κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς και η ανάλυση συνολικού κόστους. Το μεγαλύτερο χάσμα υπάρχει στο εταιρικό δίκαιο. Στη συνέχεια θα μπορούσε να μας απασχολήσει και το οικογενειακό δίκαιο που είναι πιο πολύ σχηδές και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθώς και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, έχει αποφανθεί σε ζητήματα που άπτονται του οικογενειακού δικαίου σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση και την αποφυγή διακρίσεων. Χρειάζεται λοιπόν μία εναρμονισμένη προσέγγιση. Θα προσπαθήσω να αρκεστώ στο χρόνο μου ως προς την ε, παγιοποίηση των μέσων και τη συγχώνευσή τους, ε, αυτό είναι μία επιλογή. Χρειάζεται μία κωδικοποίηση μέσα στα πλαίσια ενός συνεκτικού ε, γενικότερου πλαισίου με βάση και τη νομολογία. και ίσως χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή κωδικοποίηση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν ε, διαφορετικά ε, εθιμικά δίκαια στα κράτη-μέλη, διαφορετικό εθιμικό δίκαιο και υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης υπάρχουν ε, μερικά χάσματα γιατί δεν υπάρχει ένας πυρήνας ε, ακόμα, ο οποίος να έχει συσταθεί. Και τα όρια του που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο. Είναι δύσκολο να ενταχθούν όλα σε ένα έγγραφο, άρα η σύστασή μου βράχει και μέσο πρόθεσμα είναι να συνεχίσουμε με τη βαθμία συμπλήρωση του πλαισίου, ξεκινώντας από, το, από μη οικογενειακά ζητήματα και μετά να μας απασχολήσει το οικογενειακό δίκαιο σε σχέση με την ονοματοδοσία και την οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, ως προς την κωδικοποίηση, να δούμε πώς μπορούμε να συγχωνεύσουμε μέσα, δηλαδή ROM 1 και ROM 2, διότι θα γίνει μία αποτίμησή του στο εγγύς μέλλον και επίσης θα ήθελα να γίνει μια σωστή εφαρμογή και αποτίμηση. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο πρόεδρος, αν δούμε τα θέματα της αναγνώρισης και της εφαρμογής, βλέπουμε ότι υπάρχουν μέσα ex equator τα οποία μάλλον έχουν απαλείψει το ex equator και τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας βρίσκονται κάπου στο μέσο. Άρα θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συνεκτικό πλαίσιο ως προς την εκτελεστότητα των αποφάσεων. Και αναγνώριση των αποφάσεων. Η κατάργηση της εκτελεστότητας ξεκίνησε γιατί λέ, ε, υπόθηκε ότι έχουν ότι έχουμε άλλα εργαλεία τα οποία έχουν καταργήσει την εκτελεστότητα. Ωραία, αλλά αυτά τα εργαλεία δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν νομίζω ότι είναι καλή βάση αυτή για περαιτέρω πρόθεση νομοθεσία. Αφού κλείσουμε όλα τι τρύπε και τα παραθυράκια, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο ή ένα πραγματικό κώδικα ευρωπαϊκού α, διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Καταλαβαίνουμε ότι το πεδίο της, της θεματικής σας είναι τόσο ευρύ που ήταν ε, αδύνατο σχεδόν σε σεβαστεί το χρονοδιάγραμμα που σας δώσαμε 15 λεπτά δηλαδή. Πάμε τώρα στον ε, δόκτορα Ραντάουερ για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να κάνω μία σύντομη εισαγωγή. Έχω και στην πολιτική καινοτομία και έρευνας ε, και στις σχετικέ σχετικές μελέτες και βεβαίως θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ πέρα και ο καθηγητής Λάινελ από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ έχει όμως ανηλυμένη υποχρέωση στο Τόροντο την οποία δεν μπόρεσε να ακυρώσει. Οπότε θα τα πω εγώ. Επίσης θα ήθελα να επαναλάβω όπως είπε και η προηγούμενη ομιλητής πως ε, είναι ευρύτατο το αντικείμενο οπότε και εγώ για λεπτομέρειες θα σας παραπέμψω στο αντίστοιχο σημείο του εγγράφου. Πρώτα απ' όλα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τι είναι, γενικά είναι κάποια αποκλειστικά δικαιώματα για διάφορα πράγματα, τεχνολογικές εφευρέσεις, λογοτεχνία, ηχογραφήσεις, βίντεο, μορφές, σχήματα, χρώματα. Αλλά σημαντικό είναι να αντιληφθούμε πως δεν είναι κάτι το ενιαίο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν μιλάμε δηλαδή για εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατατεθέντα σήματα και δεν σημαίνει πάντα ότι μιλάμε για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπήρχε και από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εύρεση Τεχνιών και το, την Αρυπηρεσία την OHIM μια μελέτη η οποία έλεγε πως ε, θεωρούν όλοι οι κλάδοι πως ε, σχετίζονται σε ένα ποστό 26% με την πνευματική ιδιοκτησία ακόμα και τα άρτα της εφημερίδες ε, που διαβάζετε δείχνουν πως ε, το ζήτημα είναι σημαντικό και από οικονομική σκοπιά βεβαίως. Ταυτόχρονα τα δικαιώματα αυτά είναι ένα ζήτημα επίμαχο. Αρκετοί είναι κατά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλοι βεβαίως είναι υπέρ. Ποιος έχει δίκιο δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη και οριστική απάντηση. Άλλοι λένε πως... Ε, μάλλον το ερώτημα είναι εάν στηρίζει ή εμποδίζει την καινοτομία. Ε, η απάντηση είναι ναι και στα δύο περιέργως. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες στηρίζει και άλλες οι οποίες εμποδίζει την καινοτομία, αλλά είναι δύσκολο κάποιος να λάβει την απόφαση να το καταργήσει γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε υπό συνθήκε εργαστηρίου, παραδείγματος χάρη, τι θα γινόταν εάν δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία. Το βασικό λοιπόν είναι γιατί υπάρχει το δίκαιο αυτό. Οι υπέρμαχοι λένε πως ε, είναι με βάση κάποια άλλα φυσικά δικαιώματα, όπως παραδείγματο χάρη η ελευθερία έκφρασης ε, και έχουν πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα που οδηγούν βεβαίως σε κάποια επιχειρήματα με βάση την οικονομία, ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι χαράζουν την πολιτική πρέπει πάντα να έχουν κατά νου πως πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων αυτών που έχουν τα δικαιώματα, τα τρίτα μέρη που δεν έχουν τα δικαιώματα και βεβαίως το γενικό συμφέρον. Τώρα, ε, εδώ πέρα η εργασία μας θα ασχοληθεί με κάποια τέτοια μέσα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι λίγο πολύ γνωστά, με τα εμπορικά σήματα, με το copyright και επίσης με τα εμπορικά μυστικά. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο δεν μας απασχολεί γιατί δεν το θεωρήσαμε τόσο σημαντικό ήταν τα σχέδια. Ξεκινώντας από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αυτά στόχο έχουν να προστατεύσουν τεχνολογικές εφευρέσεις ε, που πληρούν ε, ορισμένα κριτήρια. Αυτά τα ελέγχουν ε, τα γραφεία ευρεστεχνίας δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το νέο, να έχουν ένα, ε, μια εφηβρετική εξέλιξη, να έχουν κάποια εφαρμογή στη βιομηχανία ίσως. Επίσης, κάτι το οποίο ίσως ε, είναι κάπως διαφορετικό από αυτά τα οποία γνωρίζετε είναι πως η νομοθετική δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια δεν είναι τόσο έντονη σε σχέση με άλλα μέσα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ευρεσιτεχνιών του 1970 που έφτιαξε ένα σύστημα λογικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες της βιομηχανίας. Παρά τις ε, συζητήσεις ε, για ένα ενιαίο δίπλωμα. Επίσης η Ευρωπαϊκή αυτή σύμβαση δεν ε, οδηγεί σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλλά σε απόδοση πολλών εθνικών διπλωμάτων. Έτσι στο παρελθόν είχε γίνει μια τσαπατσούλικη συζήτηση για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενώ εννοούσαμε μια εναρμονισμένη αίτηση προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και θα γινόταν μια εξέταση αλλά μετά θα έπρεπε να αποφασίσει κάποιος σε ποια χώρα θα ήθελε να ισχύει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έτσι ήταν η κατάσταση για πολύ καιρό και υπήρχαν πολλές προσπάθειες από τη δεκαετία του 1970 για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση και να καταλήξουμε σε μια πραγματικά ενιαία, σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα. Υπήρχαν ησυχίε για το γλωσσικό καθεστώς, για άλλα διοικητικά ζητήματα και κυρίως Βεβαίω το ότι κάποιοι ειδικευμένοι δικηγόροι και εθνικές υπηρεσίες στα εθνικά γραφεία ευρεσιτεχνίας ήταν κατά αλλά με το μέσο της ε, ενισχυμένης συνεργασίας 25 ε, κράτη-μέλη προχώρησαν και στην τελευταία ε, νομοθετική περίοδο είδαμε το πακέτο του ενιαίου διπλώματος με πρώτα απ' όλα τον κανονισμό 1257 του 2012 του Συμβουλίου μετά ε, το πακέτο για γλώσσες και μετάφραση και τέλος μια συμφωνία για ένα ενιαίο δικαστήριο για ζητήματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό ίσως χρειάζεται κάποια εξήγηση γιατί όταν ήταν εθνικά τα διπλώματα τότε η εφαρμογή του νόμου ήταν εθνική υπόθεση με κάποιες αρνητικές συνέπειες, δηλαδή διάλεγε κανείς σε ποιο δικαστήριο θα πάει, ή μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές χώρες. Οπότε για να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα χρειάζεται και ένα δικαστήριο με αποφάσεις για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συζητηθεί αυτά τα πράγματα. Το θέμα όμως είναι πως μόνο με τα την κύρωση της συμφωνίας από έναν ορισμένο αριθμό χωρών μεταξύ των οποίων Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία θα τεθεί ενισχύ. Οπότε αυτή τη στιγμή ακόμα και αν ο κανονισμός ο 1257 ε, του 2003 θα τεθεί ενισχύ το νωρίτερο το 2015. Και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ακριβώς να δει την εφαρμογή που θα είναι δύσκολη. Θα έχουμε συζητήσεις για τα τέλη και τις χρεώσεις ε, και βεβαίως ε, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι δημοφιλές το σύστημα γιατί μπορεί να χρησιμοποιούν και τα παλιά συστήματα και παραλλού και ίσως να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος με τα παλιά συστήματα. Τώρα, θα τα επιταχύνω γιατί έχω φάει τα δύο τρίτα του χρόνου μου. Το επόμενο εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα τα οποία βεβαίως ε, ευρεώνονται το ποιος ε, προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Στον τομέα αυτής της νομοθεσίας είχαμε δύο βασικές, ε, βασικά νομοθετήματα στο παρελθόν, η σχετική οδηγία του 98 και η οδηγία α, για το κοινοτικό εμπορικό σήμα και μια σχετική υπηρεσία όπου κατά τη είχαμε πολύ νομολογία στον τομέα αυτών για το πώς ε, πρέπει να ερμηνευθούν οι οδηγίες ε, και οι κανονισμοί και τώρα έχουμε ε, δύο νομοθετήματα που στόχο έχουν την επικαιροποίηση της νομοθεσίας. Περσινά ήταν αυτά πρόταση νομισμού που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου για τα εμπορικά σήματα και περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει τοποθετηθεί, το ίδιο και το Συμβούλιο. Το ένα θέμα στο οποίο δεν συμφωνούν αυτή την στιγμή είναι το θέμα των εξαιρέσεων. Αυτό το οποίο δηλαδή θα ήθελε να δει κάπως ε, γρήγορα το Κοινοβούλιο. Copyright κατόπιν, προστασία, εδώ πέρα μιλάμε για έργα τέχνης και ε, εδώ πέρα βλέπουμε την εξής κατάσταση. Η εναρμόνιση είναι πολύ λιγότερη από ότι με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα Και βεβαίως έχουμε μία προσέγγιση η οποία ήταν αργή και σταδιακή. Ε, πρόκειται για μία σειρά οδηγιών που εναρμόνει σε κάποιες πτυχές του σχετικού δικαίου. Πρώτα απ' όλα εστιαζόταν σε κάποιες πτυχές τεχνολογίας. Δορυφορική τεχνολογία, καλωδιακή τηλεόραση, που εκεί πέρα υπήρχαν προβλήματα με το copyright ε, και μετά υπήρχαν κάποια γενικότερα ζητήματα. Στην τελευταία νομοθετική περίοδο υπήρχαν τρεις τέτοιες οδηγίες που προσθέθηκαν στο κεκτημένο. Ε, το ένα αφορούσε ε, τροπολογία της διάρκειας της ε, ε προστασίας. Μετά υπήρχε ε, μια οδηγία για κάποια έργα π.χ. μπει σε μια βιβλιοθήκη, θέλεις να ψηφιοποιήσεις ένα βιβλίο και δεν βρίσκεις ε, τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Υπήρχε και μια οδηγία για τη συλλογική διαχείριση με στόχο ε, να ρυθμίσει την λειτουργία των εταιριών πνευματικής ιδιοκτησίας που συλλέγουν τα δικαιώματα. Αυτά ήταν λοιπόν τα ζητήματα και η Κομισιόν ξεκίνησε και κάποιους διαλόγους για άλλα ζητήματα προστασίας ε, της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και των εξαιρέσεων και αναμένεται μια λευκή βίβλος για το 2040. Τι επιφυλάσσει το μέλλον ε, πρόθεσμα αφορά πιθανώς ε, το πεδίο εφαρμογής δικαιωμάτων οδηγίες, αλλά ίσως μπορούμε να σκεφτούμε ήδη κάποιο ενιαίο ευρωπαϊκό copyright. Ήδη ομάδα έχει κάνει κάτι σχετικό για τις πιθανές κατευθύνσεις που θα μπορούσε να πάρει αυτό. Το επόμενο, εμπορικά μυστικά. Υπάρχει μια συζήτηση για το εάν συμπεριλαμβάνονται αυτά στον τίτλο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά τώρα πλέον συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία βλέπετε πως οι περισσότερες εταιρείες αποδίδουν πολύ περισσότερη σημασία στα εμπορικά μυστικά από ό,τι στην προστασία ε, των σημάτων. Ποια είναι τα εμπορικά μυστικά. Ε, δεν είναι τόσο απλό να πει κάποιος ότι κάτι είναι μυστικό. Πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια σύμφωνα με τις συμφωνίες TRIPS. Δηλαδή μιλάμε για πληροφορίες εμπορικής αξίας, οι οποίες έχουν αξία επειδή είναι μυστικές. Ε, και αν ε, ε, ισχύουν αυτά, τότε ναι, μιλάμε για εμπορικά μυστικά. Και παρέχεται κάποιο επίπεδο προστασίας. Το θέμα είναι πως ο νόμος, η νομοθεσία σχετική είναι τελείως διαφορετική από χώρα σε χώρα και δεν είναι βεβαίως ιδανική εφαρμογή σύμφωνα με την αξιολόγηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε υπάρχει μια πρόταση για Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι τώρα επιτάπητος και μάλλον θα συζητηθεί στο προσεχές μέλλον από το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αναφέρονται στο έγγραφό μας. Το ένα αφορά τη γνωστή ιστορία βεβαίως της εφαρμογής του νόμου πάντα η βιομηχανία πιέζει για να εφαρμοστεί ο νόμος. Θα υπάρξει ανακοίνωση της Κομισιόν για ένα σχέδιο δράσης για τις παραβιάσεις ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας και υπάρχει το ζήτημα των ε, διεθνών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλές συνθήκες και παραδείγματος χάρη υπάρχει ο σχετικός διεθνής οργανισμός ε, αλλά και η συμφωνία TTIP επίσης θα περιέχει κάτι για την πνευματική ιδιοκτησία. Ίσως η TTIP συμφωνία η διατλαντική ναι, εντάξει έχει ακόμα μυστικές συζητήσεις αλλά για να αντιληφθείτε την τεράστια σημασία που της αποδίδεται στις ΕΠΑ φαίνεται πως ε, πέρα από τις ε, ενδοευρωπαϊκές δραστηριότητες ε, βλέπουμε πως ο δεύτερος σημαντικότερος εταίρος μας είναι η ΕΠΑ όταν μιλάμε ακριβώς για άδεια χρήση κάποιου προστατευμένου αγαθού. Οπότε βλέπετε σε τι ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Σας ευχαριστώ. Αυτά εν περιέχει η παρουσίασή μου. Νομίζω δεν χρησιμοποίησα πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε για τη γρήγορη επισκόπηση του θέματος ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δυστυχώς θα αναγκαστώ να φύγω από την ακρόαση και θα ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο, την κυρία Ντελβό, να προεδρεύσει τη θέση μου. Έχω ένα ραντεβού. Ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ για την συνεισφορά σας. Μέχρι εδώ μπόρεσα να ακούσω, μέχρι εδώ θα μπορέσω να ακούσω, ζητώ συγγνώμη. Θα περάσουμε απευθείας στην τελευταία παρέμβαση και θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Παλμερίνη και στον ε, καθηγητή Μπερτολίνη we share presentation. <laughs> Thank you and Θέλω να σε ευχαριστήσω που μας καλέσατε και μας δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε για την έρευνα που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Um, Η ρομποτική είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που θα μετασχηματίσει εκβάθρον την κοινωνία μας. Ε, επενδύονται τρομερές, τρομερα, τρομεροί πόροι, ε, περνάνε νόμοι σχετικά, ούτω ώστε να προωθήσουμε την ρομποτική, το ρομποτικό κλάδο, τα ΜΜΕ και άλλα μέσα ε, ενδιαφέρονται και αναμένεται τεράστια οικονομική επίπτωση από την ε, πρόθεση της ρομποτικής στις υπηρεσίες, ε, στον τομέα της υγείας, ε, λοιπά. Μόνο στον τομέα της υγείας θεωρούμε ότι τεχνολογίες όπως ε, τα προσθετικά, εξωσκελετικά, ε, χειρουργική με ρομπότ, ε, βοήθεια για ηλικιωμένους μπορεί να βελτιώσει τρομερά τη ζωή και να παρατείνει τη ζωή των ανθρώπων. Ε, αυτόνομα οχήματα επίσης μπορεί να μειώσουν τα ατυχήματα και να σώσουν ζωές. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να εντοπίσουμε την ε, ρομποτική ως ένα μείζον θέμα που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγύψει από αυτού, τόσο ώστε να γίνει παγκόσμιος παίχτης και να προωθήσει και τις δημοκρατικές αξίες μέσω αυτής. Η τεχνολογία της ρομποτικής είναι και ευκαιρίες, αλλά για να είμαστε έτοιμοι για τις ε, προκλήσεις αυτού του νέου κλάδου θα πρέπει να έχουμε ε, ένα νομικό σώμα, ένα ε, ρυθμιστικό κανονιστικό περιβάλλον ε, κατάλληλο, διαφανές, να ξέρουμε ότι οι προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να τεσταριστούν και συνεχεία να δρομολογηθούν στην αγορά. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία, να μην δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη υψηλών, ε, υψηλής τεχνολογίας, όπως φοβόμαστε, αντίθετα να εκμεταλλευτούμε το τεράστιο δυναμικό της ρομποτικής. Για να είναι όμως μια τεράστια ευκαιρία η ρομποτική θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με την ε, ιδέα της ε, υπεύθυνη έρευνας και καινοτομίας και να υπάρχει συνάφεια με τις θεμελιώδεις αρχές που όπως εγγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ενωμή Τάξη. Μία παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται από την, το διασυναριακό χαρακτήρα της έρευνας που γίνεται στον τομέα αυτό και από την τεχνολογική καινοτομία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνεργασίας διαφόρων ερευνητικών ομάδων ε, που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες. Θα πρέπει να έχουμε πόρους και ρυθμιστικά εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη τη διασυνορική διάσταση του κλάδου. Ε, ηθική αποδοχή, ε, προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες ε, για να έχουμε την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. Τα ρομποτικά προϊόντα και εφαρμογές θα πρέπει να συμμορφούνται με τις βασικές αξίες της Ευρώπης, αλλά θα πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμογές αυτές που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και επομένως συνεισφέρουν στην υλοποίηση στόχων όπως ε, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ίσες ευκαιρίες. Αυτή η τεχνολογία θα πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ε, ειδικά των πιο ευπαθών ομάδων και μπορεί να προωθηθεί μέσω της υιοθέτηση κατάλληλων νομοθετικών ε, μέτρων. Το πρόγραμμα Ρομπόλο που συντονίζω έχει σκοπό να δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βασική έμπνευση είναι να δώσουμε στους ερευνητές κοινωνικές αξίες και διοντολογία για να τις ενσωματώσουν στην έρευνα. Οι επιλογές επίπεδο πολιτικής απαιτούνται ήδη με την με το επίπεδο, λόγω του επίπεδου που έχει φτάσει η τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που είναι γενείς στη ρομποτική. Μιλάμε για τεχνολογίες προσθετικής που προωθούνται μέσω της ρομποτικής και που ε, συμπληρώνουν ακροτηριασμένα μέλη κτλ. Και μπορεί να προσθέσουν και νέες λειτουργίες ε, στο ανθρώπινο σώμα που τις έχει χάσει ή δεν τις έχει. Αντί να χρησιμοποιούμε με θεραπευτικό μόνο τρόπο τη ρομποτική τεχνολογία, αλλά αν τη χρησιμοποιούμε ε, ως ενίσχυση των ε, των ικανοτήτων του ανθρώπου ε, μας κάνει να σκεφτόμαστε για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, για τα όρια στις δυνατότητες ε, αύξηση των ικανοτήτων μας. Θα αντικαταστήσουμε, παραδείγματο χάρη, ένα υγιές ε, σώμα, ε, ένα υγιές μέλος με ένα βιονικό γιατί θα μας βοηθήσει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα. Μπορεί να έχουμε τρομακτικά παραδείγματα, γιατί η ενίσχυση των ικανοτήτων μας μέσω της ρομποτικής μπορεί να επηρεάσει πολλά, πολλές ικανότητες. Ε, την ενίσχυσή μας, την ικανότητα μας να μαθαίνουμε ακόμα, ε, τη, τη ταχύτητα κτλ. Μπορεί να έχουμε και καθαρά χρηστική λειτουργία Ε, και ο σκοπός είναι το μέγιστο, η μέγιστη ευημερία του συνόλου. Αλλά δεν πρέπει να το δούμε μόνο έτσι. Γιατί οι αρρώστιες, ε, η εξάρτηση που θέλουμε να ξεπεράσουμε ε, αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστές στην κοινωνία μας. Και ορισμένοι θεωρούν ε, ότι αυτές οι ασθένειες, οι αδυναμίες μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αν τέτοιες ε, τεχνολογίες όμως ε, μπορούν να μειώσουν τις αναπηρίες και τις, ε, τις αδυναμίες, μπορούν να δημιουργήσουν νέες, νέα προβλήματα, δηλαδή εξάρτηση πια από την τεχνολογία. Μία νομική κατανόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη λοιπόν, καταρχάς για να εξασφαλίσουμε την συνάφεια με το συνταγματικό κοινό πλαίσιο και με την αρχή της προφύλαξης, όπως ε, αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους επιστήμονες. Υπάρχουν όμως και άλλοι πιο ρεαλιστικοί λόγοι ε, που μας οδηγούν στην υιοθέτηση κοινή τάση απέναντι σε αυτό το θέμα και να μην το αφήσουμε απλώς σε μια πολυσχηδή αντιμετώπιση των κρατών μελών. Δηλαδή, ε, αν έχουμε διάφορες νομοθεσίες μπορεί να επηρεάσει την, κινήση, την κινητικότητα μάλλον διαφορών υπηρεσιών και αγαθών. αυτό το βλέπουμε σε άλλους τομείς, σε άλλα βιο δεοντολογικά βιοειθικά σενάρια και να οδηγηθούμε σε ανταγωνισμό μεταξύ νομικών συστημάτων. Χρειαζόμαστε να έχουμε διασυνοριακούς κανονισμού, ώστε να αποφύγουμε τέτοιους περιορισμούς και απαγόρευση σε κάποιες χώρες. Ε, και να μην υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ χωρών ε, ανάμεσα σε αυτές που επιτρέπουν πιο πολύ και σε αυτές που περιορίζουν. Μπορούμε να υποστηρίξουμε και τι εθνικέ αποφάσει σε κανονιστικό επίπεδο ε, για τους νομοθέτες, αλλά και σε πιο πρακτικό επίπεδο, το χάρη, στα οι φορείς υγείας, όταν χρειάζεται να αποφασίσουν για μια παρέμβαση, ας πούμε, ε, αναπερίπτωση, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ο συνάδελφός μου θα συνεχίσει την παρέμβασή μου. Πριν ε, μιλήσουμε για την ρύθμιση της ρομποτικής θα πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Η λέξη αυτή αναφέρεται σε κάτι που μοιάζει με άνθρωπο που περπατά ή μιλάει. Αλλά αν δείτε τις εικόνες βλέπετε τις διαδικασίες προσθετικής Επίσης βλέπετε ένα ρομπότ το οποίο καν δεν διαθέτει ε, σώμα και δίνει απαντήσεις και υπάρχει και ένα χειρουργικό ρομπότ ε, το οποίο ελέγχεται από μία κονσόλα και επίσης ένα μη επανδρομένο όχημα και επίσης ε, κάτι που μοιάζει με τον ορισμό που δώσαμε, δηλαδή ε, ένα συγκεκριμένο ρομπότ για την αποκομιδή, το οποίο φτιάξαμε στην Πίζα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία καταπροσέγγιση περίπτωση και να μην έχουμε έναν ενιαίο ε, κώδικα που να διέπει τη ρομποτική. Θα πρέπει να έχουμε μία αναπερίπτωση προσέγγιση Επίσης, μάλλον ε, οι ίδιες τεχνολογικές ε, ε, τάσεις δεν σημαίνουν εν ενίο πλαίσιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μία αυτόνομη ηλεκτρική σκούπα έχει ε, ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας από ένα μη επανδρομένο όχημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι επιπτώσεις αυτής της τεχνολογίας στην κοινωνία. Δεν φαίνεται αυτή η διαφάνεια. Και το ίδιο νομικό ζήτημα ίσως χρειάζεται διαφορετικές ε, λύσεις ε, Δηλαδή, αν μιλάμε για την ε, προσθετική με βάση τη ρομποτική και ένα ε, μη επανδρομένο όχημα και μιλήσουμε για την ευθύνη σε περίπτωση ζημίας, το θέμα είναι πολύ διαφορετικό, διότι αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε τα σωστά κίνητρα ανάλογα με την συγκεκριμένη εφαρμογή και κατά πόσο είναι επιθυμητή θα ήθελα εντάχει να δούμε τα ζητήματα κατανομής ευθυνών. Ε, ευθύνη σημαίνει ποιος θα καταβάλει το αντίτιμο, την αποζημίωση δηλαδή σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας. Γιατί υπάρχει ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως το ίδιο το ρομπότ ίσως φέρει την ευθύνη. Αυτό φαίνεται παράλογο, αλλά ισχύει όπως ισχύει και σε, και στη, σε μια κοινοπραξία, δηλαδή στη, σε μια καθαρά εταιρική βάση. Ποιοι είναι οι, οι στόχοι των κανόνων ε, ευθύνης αφορά ένα κοινό νομικό ε, πλαίσιο που διέπει το καθεστώς αποζημιώσεων. Αν πρόκειται για ένα προϊόν ε, το οποίο ε, ένα προϊόν το οποίο είναι ελαττωματικό θα πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ποιος ε, φέρει την ευθύνη. Ε, και το, σε περίπτωση μη επανδρομένου οχήματος, αυτό μας ενδιαφέρει είναι σε περίπτωση ατυχήματος ποιος φέρει την ευθύνη, ο κατασκευαστής, ε, τη στιγμή που δεν υπάρχει οδηγός. Και αυτό αφορά και την οδηγία ελαττωματικών προϊόντων. Η οδηγία ελαττωματικών προϊόντων, για τα ελαττωματικά προϊόντα, ε, μιλά για επιπτώσεις που φυσικά δεν είναι επιθυμητές. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά 97% τα ατυχήματα σε αιτήσια βάση με βάση τη ρομποτική. Τι γίνεται ως προς την, ε, το καθεστώς αποζημιώσεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ασφαλιστικά συστήματα με συμβαλόμενο και αντισυμβαλόμενο μπορείτε να διαβάσετε τα συμπεράσματα στο έγγραφο σε σχέση με την ε, προσθετική και ένα πρόσθετο ε, μέλος. Ένα ρομποτικό χέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς λόγους, για οδήγηση, και για να κρατά μια τσάντα με ψώνια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο ε, υπάρχει σοβαρή περίπτωση ατυχήματος. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τις συνέπειες και πολλές φορές ε, είναι πολύ δύσκολο να ε, καταχωρήσουμε το λάτωμα. Το άρθρο 4 των, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ΑΜΕΑ ορίζει τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και συγκεκριμένους νόμους περί ευθύνης. Πώς ορίζονται αυτοί οι νόμοι περί ευθύνης. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ορισμένες εξαιρέσεις για τους κατασκευαστές. Όταν πρόκειται για χειρουργικά ρομπότ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ υπάρχει και ο χειρούργος ε, και το μηχάνημα. Εδώ υπάρχει ε, ένας διαφορετικός επιμερισμός ευθυνών και πολλές, πολλές φορές ίσως υπάρχει αμέλεια θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την κατανομή αυτών των ευθυνών. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποδώσουμε την ευθύνη στον κατασκευαστή και όχι στον χειρουργό. Σε πολλές περιπτώσεις ίσως θα πρέπει να περιορίσουμε τη δράση μας ε, και σε περίπτωση προσφυγής θα πρέπει ο ασθενής να γνωρίζει τις πληροφορίες ε, χρήσης. Επίσης, ως προς την προσωπική φροντίδα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ύπαρξη ενός ρομπότ για ε, ανθρώπους ε, προχωρημένης ηλικίας, για ηλικιωμένους ή για χρήση από ανθρώπους με κινητικά και άλλα προβλήματα. Εδώ ε, συζητάμε κατά πόσο θέλουμε να μιλήσουμε για μία νομική οντότητα δεν μπορεί να φέρει ευθύνη το ρομπότ όπως ε, φέρει μια εταιρεία για παράδειγμα. Γιατί ε, γίνεται χρηματοδότηση είτε από τον κατασκευαστή είτε από το χρήστη έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνης. Ε, ως προς τα ρομπότ προσωπικής ε, φροντίδας θα βοηθούσαν ιδιαίτερα ε, του ηλικιωμένου ή τους ανθρώπους με κινητικά και άλλα προβλήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιο είναι το μακροχρόνιο ε, κόστος και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η περίπτωση αποζημίωσης. Αν θέλουμε να δούμε ε, τα προϊόντα από πλευράς ασφάλειας. Υπάρχουν κάποιες εμπειρικές μελέτες που δείχνουν πως δεν παρέχονται εδώ πέρα περαιτέρω κίνητρα. Οι περισσότεροι κανονισμοί ασφαλείας στην Ευρώπη είναι κάποιες οδηγίες που έχουν ευρύτατο πεδίο εφαρμογής. Π.χ. αν πάρετε τα ενεργά εμφυτεύματα, τα ιατρικά, είναι τα πάντα από βηματοδότη μέχρι τεχνητό χέρι που και διαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Επίσης, αν μιλάμε για ιατρικά εργαλεία, μιλάμε για ε, ιατρικά γάντια μέχρι έναν εξωσκελετό που είναι ένα ολόκληρο ρομπότ. Οπότε υπάρχει και ο ο οργανισμός ε, και θα πρέπει να πάμε σε πιο στενές τεχνικές προδιαγραφές ε, οι οποίες θα είναι αρκετά υψηλές και θα πρέπει να τηρούν η παραγωγή επίσης θα πρέπει να δούμε και τις επαγγελματικές απαιτήσεις παραδείγματος χάρη η γη οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά. Ένα σύστημα δηλαδή αδειοδότησης. Ήδη υπάρχουν κάποιες μελέτες ε, στη ΣΥΠΑ και πρέπει να συμπληρώσουμε το κενό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά και για να ολοκληρώσουμε οι σκέψεις αυτές ε, τις οποίες ανέπτυξα αναφέρονται και στο έγγραφό μας ε, και σε ένα έγγραφο το οποίο εκδώσαμε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση των, ε, της ρομποτικής και εκεί πέρα προσπαθούμε να αναλύσουμε με λεπτομέρεια τις τεχνολογίες αυτές, τα προβλήματα που παρουσιάζουν και προτείνουμε κάποιες ε, πολύ συγκεκριμένες ε, τεχνικές λύσεις που θα μπορούσαν ήδη να χρησιμοποιηθούν εάν υπήρχε η πρόθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την εντυπωσιακή αυτή παρουσίαση. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. 15 λεπτά. Η κυρία Ρέιντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ειδικού. Έχω μία ερώτηση για το copyright και μία για την ομοθεσία περί ρομποτικής. Για το copyright, ε, κύριε Ράντο, στις ε, πρόσφατες ε, διαβουλεύσεις πολλοί από τους τελικούς χρήστες ρωτούσαν συγκεκριμένα για κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην καθημερινή του ζωή. Το ένα αναφέρει το πρόβλημα διασυνοριακής ε, πρόσβασης ε, σε περιεχόμενο το οποίο νομίμως έχουν ε, στο διαδίκτυο και αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό διασυνοριακά και για τα ρομπότ. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια συζήτηση όχι μόνο για την ευθύνη αλλά και από την πλευρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί, όπως εξηγήσατε και στα τεχνητά μέλη, υπάρχει βεβαίως το θεμελιώδες δικαίωμα της σωματικής ακαιρεότητας, το οποίο αφορά φυσικά μέλη, οπότε το νομικό όριο για το κράτος είναι πολύ υψηλότερο από ότι ε, στο να δεσμεύσει παραδείγματο χάρη ε, κάτι το οποίο είναι απλά ιδιοκτησία μου. Δηλαδή, αν θεωρείτε πως θα πρέπει να διευρυνθεί το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα ως προς αυτό. Μάλιστα. Κυρία Μολπάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν δεινόσαυρος ε, αισθάνομαι μετά την παρουσίαση για τα ρομπότ. Ε, εμένα η ειδικότητά μου είναι το ποινικό και το οικογενειακό δίκαιο και η ρομαντική μου αν θέλετε ερώτηση είναι μια που διάβασα και το έγγραφο ε, βλέπουμε ε, πως λέτε πως μπορεί να πάνε οι ευθύνες φροντίδας στα ρομπότ, να ανατεθούν σε ρομπότ. Ε, δηλαδή η αγάπη και η φροντίδα για τον ηλικιωμένο, όλα αυτά τα ρομαντικά πράγματα θα πάνε στα ρομπότ. Και αυτά τα οποία λέγαμε, η γονεϊκή ευθύνη, η ευθύνη του παιδιού απέναντι στον ηλικιωμένο γονέα, τον άρρωστο συγγενή, πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά. Τι, εγώ θα αφήσω τη μάνα μου με ρομπότ. Θα ήθελα Τα σκέφτεστε αυτά ή είναι έτσι πράγματα παλιωμοδίτικα και έννοιες ξεπερασμένες. Ε, τέλος. Μια που εγώ δεν είμαι έτσι πολύ των τεχνολογικών, αν μπορείτε να μου εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ ενός ε, ε, αυτοκινήτου το οποίο οδηγεί ο υπολογιστής ή κάποιο άλλο τέτοιο οχήματο. Ποια η διαφορά και αυτού από έναν υπολογιστή. Και μια ερώτηση από τα παλιά, όταν υπήρχαν γονείς, με πραγματικοί γονείς, με πραγματικά παιδιά ε, και ζούσαν σε διαφορετικές χώρες. Ε, μια χαρακτηριστική ερώτηση ήταν πως πολλοί από εμά ε, λαμβάνουμε επιστολές ε, στις οποίες ε, το όλο ζήτημα του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου και της απαγωγής παιδιών συνεχώς προκύπτει. Εάν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες οδηγίες, πρώτα απ' όλα για το ποιοι είναι οι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, όσον αφορά την απαγωγή παιδιών. Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό site ε, για την ομολογία της Σύμβασης της Χάγης, ε, το οποίο χρησιμοποιούμε. Αλλά επειδή είμαι ειδικό στον τομέα, εγώ παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνω το πώς κατησχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο του εθνικού, εάν ε, ισχύει η πρωτοκαθεδρία της Σύμβασης Χάγης κτλ. Αν μπορείτε λίγο να μου το εξηγήσετε όλα αυτά τα σημεία που αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ. Επόμενη και τελευταία ερώτηση. Κύριος Κιώστερ, το ερώτημά μου αναφέρεται στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίες. Σας ευχαριστώ πράγματι για τις πολύ καλές παρουσιάσεις σας. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα έχει κάποια επίδραση στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και αν είναι πια. Σαφής και σύντομη ερώτηση. Μπράβο. Οπότε θα δώσω τον λόγο στους ειδικού μας. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον δόκτορα Κράμερ. την Κράμερ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ πολύπλοκη η ερώτησή σας. Δεν μπορώ έτσι να σας παραπέμψω σε μία πηγή. Η σύμβαση της ε, Χάγης και η σχετική διάσκεψη ε, είναι πάρα πολύ δραστήρια. Υπάρχουν στο site πάρα πολλά πράγματα, τεκμηρίωση και βεβαίως παρακολουθούν και το τι συμβαίνει με την επιστροφή του παιδιού. Ένα άλλο ζήτημα είναι η αξιολόγηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α ε, για την απαγωγή και την επιστροφή του παιδιού που ακόμα βεβαίως ε, εξαρτάται από μια διαταγή περί του εκτελεστέου αλλά Ε, εδώ πέρα υπάρχει μια συνεργασία παραδείγματος χάρη ε, στην συνθήκη της Χάγης για κάποιες απαιτήσεις ε, που πρέπει και κάποιους όρους που πρέπει να πληρούνται. Γίνεται λοιπόν όπως είπα κάποιες σχετικές αναφορές όταν μιλάμε για την εκτροφή του παιδιού. Υπάρχει λοιπόν ε, κάποια, ε, έτσι θα έλεγα, συνεργασία. Αλλά είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Εγώ ξέρω πως υπάρχει ήδη κάποια δουλειά που γίνεται για κάποια αναθεώρηση για να υπάρχει μια αυτόματη επιστροφή του παιδιού χωρίς να κοιτάμε ε, πού και τι και πώς ή μήπως θα έπρεπε να πάμε στην κατεύθυνση όχι άμεσης επιστροφής αλλά να δούμε περισσότερο τα συμφέροντα του παιδιού. Μα είναι θεμελιώδης αυτή η συζήτηση. Δηλαδή άμα ξεκινάτε με το να λέτε πραγματικοί γονείς και πραγματικά παιδιά τι εννοούμε. Τους βιολογικούς γονείς. Νομικά. Τι. Δηλαδή τι, τι είπα να πει πραγματικός γονιός. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ε, βιολογικός γονέας, αλλά έχει κάποια σημασία στο νόμο. Αλλά ένα παιδί το οποίο είναι υιοθετημένο ή έχει αναγνωριστεί από κάποιον ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός γονιός, ε, και αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα. Ε, οπότε το θέμα είναι πράγματι ποιος είναι ο κηδεμόνας, ποιος είναι ο γονιός σύμφωνα με τον νόμο εντάξει αυτό αναγνωρίζουμε ως ε, ε, νόμιμο, αλλά τώρα δεν μπορώ έτσι γρήγορα να σας εξηγήσω ολόκληρη την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ο δόκτωρας Ραντάουερ ίσως μπορεί να μας απαντήσει έτσι σύντομα. Δύο ερωτήματα. Ένα για το copyright και τις δυνατότητες για να υπάρξει διασυνοριακή πρόσβαση στο νομίμως κατεχόμενο περιεχόμενο. Λοιπόν, για την πρώτη αυτή ερώτηση δεν είμαι νομικός, οπότε δεν μπορώ εγώ να σας πω πως είναι το άρθρο τάδε εδάφιο δίνα, αλλά μπορώ να σας πω ε, την ανάλυση του καθηγητή Χούγκεν Χόρτς για την εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου η οποία έχει ως εξής παρά το ότι οι 7 αυτές οδηγίες έχουν πλέον αμβλύνει κάποιες διαφορές ο εδαφικός χαρακτήρας ε, της σχετικής νομοθεσίας ε, παραμένει άθικτος. Αυτό σημαίνει πως η παραγωγή περιεχομένου πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα δικαιώματα σε 25 ε, περίπου κράτη-μέλη. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ε, σαφές ε, μειονέκτημα σε σύγκριση παραδείγματος χάρη με τις Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά και η απάντηση όσον αφορά το copyright. Τώρα για τη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου είναι δύσκολο να απαντήσω γιατί οι διαπραγματεύσεις για την TTIP, ε, την συμφωνία τη Διατλαντική είναι μυστικές, δεν ξέρω τι συζητάνε, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Αλλά κάποια σχόλια ίσως. Οι ΙΠΑ έχουν έναν κώδικα πρακτικής, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς, ε, ένα τριψήφιο κώδικα το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών εκεί πέρα το οποίο περιγράφει το πώς ε, ε, πρέπει να κινούνται οι διαπραγματευτές ε, των ΗΠΑ όταν μιλάνε για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Και ίσως είναι καλή ιδέα να το δούμε αυτό. Συνήθως αναφέρεται πάρα πολύ έντονα η πνευματική ιδιοκτησία, ειδικά με τις ΗΠΑ καθώς ενδιαφέρονται για να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας της πνευματική ιδιοκτησίας και συχνά αυτό γίνεται μέσω ενός πολύ συγκεκριμένου καταλόγου πραγμάτων που θέλουν να δουν και έτσι κάνουν το lobbying που κάνουν. Και λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό από πλευράς ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία και να δούμε το τι γίνεται με αυτό. Και κοιτάξτε το αν δεν το έχετε δει. Η άλλη πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω και το είπα ήδη ήταν ότι πρέπει να αντιληφθούμε την συμφωνία της Αμερικανικής αγοράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια υπόθεση που λέει πως εάν τελειώσουν αυτά και τα ζητήματα και τα φτιάξουμε στην Ευρώπη ε, διορθώνουμε το πρόβλημα. Ίσως ένα 50% του προβλήματος γιατί το άλλο 50% είναι η ΙΠΑ. Οπότε πρέπει να δούμε ε, πώς προχωράει η νομοθεσία, στη ΣΥΠΑ και το τι σημαίνει αυτό για ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν, ε, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις με την πνευματική ιδιοκτησία. Ένα 80% θα έλεγα χοντρικά όλων των σχετικών δικών ε, λαμβάνουν χώρα στη ΣΥΠΑ. Οπότε αυτό και πάλι μας λέει πως πρέπει να δούμε ε, την κατάσταση στη ΣΥΠΑ και όχι μόνο στην Ευρώπη. Ωραία, ευχαριστώ. επόμενη. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. θεμελιώδη δικαιώματα και τα μέλη. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα τεχνητά μέλη πράγματι υπάρχει εδώ πέρα ένας... Ναι. Μια επανάσταση για το σώμα. Ε, τα βιονικά εμφυτεύματα μπορούν να, ε, να προστεθούν στο σώμα, να κολλήσουν και επομένως ε, μπορεί να την αντιμετωπίσουμε ως ε, μέλη του σώματος. Ε, χάρη στο το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα στη σημαντική ακαιρεότητα μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτά τα εξαρτήματα. Και το, το καθεστώς που ισχύει στα μέλη του σώματος μπορεί να ισχύσει και στα τεχνητά μέλη. Ε, υπάρχει τέτοια νομολογία. Ε, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν είναι επίμαχο το θέμα, εντός και εκτός του δικαστηρίου. Ένα άλλο ερώτημα για την... για τα, τα ρομπότ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τους ηλικιωμένου, για την φροντίδα των παιδιών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό διοντολογικό θέμα αυτό. Το αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της έρευνά μας και είναι και το πιο ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Η ιδέα είναι ότι τα ρομπότ που φροντίζουν αναλαμβάνουν τα βαριά, τα δύσκολα καθήκοντα και απελευθερώνουν τους ανθρώπους που φροντίζουν και αυτοί για να συνεχίσουν να κρατούν συντροφιά, να μιλούν, να αγαπούν. those χωρίς να ασχολούνται με τα βαριά καθήκοντα, το πλήσιμο ας πούμε, τη φροντίδα ας πούμε, τη σωματική κτλ. Αυτό είναι ο ρόλος τεχνολογίας. Το άλλο σας ερώτημα για τα αυτόνομα οχήματα χωρίς οδηγούς. Υπάρχουν τέτοιες τεχνολογίες αυτοματοποιημένες τεχνολογίες. Είναι θέμα βαθμού καταρχήν αυτοματοποίησης. Εδώ μιλάμε για πλήρη, πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα, τα οποία οδηγούνται χωρίς ανθρώπινη εποπτεία. Ενώ στα άλλα συστήματα πρέπει να υπάρχει κάποια εποπτεία από ανθρώπους. Και μια άλλη διαφορά είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους ενώ άλλα είδη τεχνολογίας είναι τμήμα μιας υποδομής η οποία δημιουργείται για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, ε, σχεδιάζεται ειδικά δηλαδή για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ο Ανδρέα θέλει να προσθέσει κάτι. Έχω δύο νομικά θέματα, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προσθέσω κάτι. Να τονίσω ότι στην Ιρλανδία ξεκαθαρίσαμε ότι τα ρομποτικά εμφυτεύματα πρέπει να θεωρούνται τμήμα του ανθρώπινου σώματος. Για λόγους, ας πούμε, ταυτότητας. Ο Νίελ Χάρμπινσον, ας πούμε, είχε φοβερά προβλήματα ε, με, την, ε, με τις φωτογραφίες ταυτότητας, ας πούμε, όταν, φοράει, όταν φορούσε αυτά τα, τα ειδικά γυαλιά, ας πούμε, στα μάτια του, ε, πρέπει να θεωρούνται αυτά τα τμήματα της τεχνολογίας ως τμήμα του σώματος. Τώρα, για το θέμα της φροντίδας με ρομπότ, ε, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες, με ανάπηρους κτλ. Και, και μας λένε ότι ο χρόνος που ξοδεύουμε ανθρώπους είναι χρόνος που καταναλώνεται ας πούμε, για να τους φροντίσουμε βαριά καθήκοντα και δεν έχουν λόγω αυτής της, της πατάλης στα βασικά, σε βασικές ανάγκες δεν έχουν χρόνο να έχουν πραγματική συζήτηση, να ε, κάνουν παρέα σαν άνθρωποι ας πούμε. Ο άνθρωπος, ο, άνθρωπος ο οποίος ξοδεύει το χρόνο του για να ταΐσει έναν ανάπηρο ε, αντί να τον τάσει, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει συζήτηση και το τάισμα το κάνει το κομπιούτερ, το ρομπότ. Ε, και αισθάνονται αυτοί οι ανάπηροι ε, πιο περιθωριοποιημένοι εξαιτία αυτή τη αντιμετώπιση. Ε, και αυτό μας το λένε διάφορες ομάδες ε, οι οποίες, με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια των ε, ερευνητικών μας προγραμμάτων. Άλλες ερωτήσεις? σύντομα. C-175 είναι η αντίστοιχη διαδικασία των Αμερικανών. Είναι άλλη συμφωνία από τη Συμφωνία Ελευθέρου ε, Εμπορίου. Μοιάζουν με τις ε, συμφωνίες ε, C-175 Ελευθέρου Εμπορίου βέβαια. C-175. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους εμπειρογνώμονες για την πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή τους, παρεμβάσεις τους, συμμετοχή τους και όλους σας. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το εργαστήρι. Θα ήθελα να το επαναλάβουμε σύντομα. Ευχαριστώ.